Uh, uh, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλέσω να καθίσετε. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την τόσο σημαντική συζήτησή μας για την οδηγία για το δικαιώμα των καταναλωτών. Good. Well, can I, um- Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω όλους θερμά στην σημερινή απογευματινή συζήτηση για την οδηγία για το δικαίωμα των καταναλωτών. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Αντρέα Σφάμπο, που κάθεται εδώ στα αριστερά μου και ο οποίο είναι ο εισηγητή τη πρόταση. Διότι, τον ευχαριστώ διότι ε, είναι ο βασικό υπεύθυνο μαζί με τη Γραμματεία για την οργάνωση αυτή τη ακρόαση. Δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Τον πιέσαμε κατά κάποιο τρόπο γιατί σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τρέχοντας με την πρόταση αυτή. Είμαστε, είμαστε λοιπόν, συμπειρογνώμονες που ήρθαν. Δεν τους ε, παρουσιάσω έναν ένα σε αυτό το στάδιο. Έχετε την ημερήσια διάταξη μπροστά σας. Στόχος είναι να μείνουμε τόσο των χρονικών πλαισίων στο βαθμό που γίνεται βέβαια κάτι τέτοιο ζητώ από όλου του ε, προσκεκλημένου μα να προσπαθήσουν να μείνουμε στα περιθώρια χρόνου που έχουν στη διάθεσή του, γιατί είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει. Θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα την κυρία Πάολα Τεστόρη Γκότσι, η οποία είναι υποδιευθύντρια τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, ε, η αναπληρωτήρια διευθύντρια, και την ευχαριστώ διότι ε, μας έδωσε ε, το πολύ σημαντικό συμπληρωματικό έγγραφο το οποίο κατάρτισε η Επιτροπή. Ε, ε, δύο μάλλον. Το ένα ξεκαθαρίζει την ε, πρόταση και το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό έγγραφο και είναι ένας πίνακας με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις διάφορες χώρες. Κάτι το οποίο θέλουμε να ζητήσουμε εδώ και καιρό. Και οι εμπειρογνωμονές μας νομίζω θα χαίρονται ιδιαίτερα με το έγγραφο αυτό. Ε, και θα σας πω, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν, η σημερινή ακρόαση, στην ουσία, αποτελεί την αρχή του νέου σταδίου της αναθεώρησης της ακμέρους ε, Επιτροπής μας ε, της ε, οδηγίας αυτής. Κάτω από την έμπειρη καθοδήγηση της προκατόχου μου, της κυρίας Μακάρθη, ε, η Επιτροπή έκανε ε, πολύ σημαντική εργασία αναλύοντας την ε, πρόταση, εξετάζοντας την αξιολόγηση αντίκτυπου και είχαμε και τότε μία ακρόαση εμπειρογνωμόνων για να ενημερωθούμε. Τώρα χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχουμε ένα εισηγητή, τον Άντρε Σβάμπ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα καταρτισμένος για να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Έχουμε επίσης ε, ε, και μια ισχυρή ομάδα σκιωδών εισηγητών και τώρα αυτό που θέλουμε είναι να ασχοληθούμε με το νομοθετικό έργο, να προτείνουμε τροπολογίες και να προχωρήσουμε στην νομοθετική διαδικασία. Αυτή λοιπόν είναι η κρίσιμη αναρτήρια συζήτηση τη όλη διαδικασία. Χωρί καθυστέρηση λοιπόν, να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον Άντρια Σβάμπου, για να κάνει κάποιε προκαταρκτικέ παρατηρήσει και στη συνέχεια θα προβούμε ε, στην ε, ακρόαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ε, λίγο περίεργο για μένα που κάθομαι εδώ μαζί με το Προεδρείο σήμερα, αν και δεν είναι ε, περίεργο για μένα που κάθομαι δίπλα σου, Μάρκο. με πάση περιπτώσει, ε, χαίρομαι για αυτή την ακρόαση που οργανώνουμε σε ό,τι αφορά αυτή την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή και ελπίζω πως οι εμπειρογνώμονες που έχουμε σήμερα εδώ θα μας βοηθήσουν τη συζήτηση και χαίρομαι με το γεγονό ότι το πάνελ αυτό είναι τόσο μεγάλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συνεργάτε εδώ ε, τη Γραμματεία, ειδικότερα την κυρία Μπαρόν, για την προετοιμασία τη σημερινή ακρόαση. Ε, τα έβραξαν αυτά πολύ καλά. Και εγώ συζήτησα με εισηγητέ από άλλε πολιτικέ ε, ομάδε, οι οποίοι ήταν όλοι του διατεθειμένοι να διοργανώσουμε αυτή την ακρόαση, ακόμα και αν ήταν ασφιχτό το χρονοδιάγραμμα, η κυρία και Τριανταφυλλίδης ήταν οι συνάδελφοι λοιπόν που συνεργάστηκαν μαζί μου και νομίζω ε, πως με αυτή τη βάση ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με την απαραίτητη επιμονή αλλά και δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στον εαυτό μας ούτως ώστε αυτή η πρόταση και αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό για τα δικαιώματα του καταναλωτή να εξεταστεί με το σωστό τρόπο και με το χρόνο που χρειαζόμαστε. Γιατί βέβαια θα πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ αφενός ε, μιας ε, προσφοράς ε, προϊόντων για τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά που θα είναι υψηλή ποιότητα, αλλά ταυτόχρονα και προστασία των καταναλωτών αφετέρου. Εάν προσπαθήσουμε και αν καταφέρουμε να βρούμε τη χρυσή τομή εδώ, θα έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Άρα λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ε, διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, αλλά με το γεγονό ότι θα πρέπει οι καταναλωτέ και επιθυμούν να έχουν μια ευρία ποικιλία και καλέ ε, τιμέ, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να καταβάλουν ένα μέρο ε, τη μεγαλύτερη αυτή νομική προστασία τη οποία θα νομίζω πως ε, θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστο εάν, για παράδειγμα, έχουμε ε, μείωση κάποιων διαδικαστικών δαπανών σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Καθώ μέχρι στιγμή στα 27 διαφορετικά κράτη-μέλη είχαμε 27 διαφορετικά συστήματα τα οποία ίσια. Αν λοιπόν επιτύχουμε κάτι τέτοιο εδώ και έχουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά, τότε νομίζω πω θα έχουμε ε, επιτύχει με καλύτερο τρόπο στην ασφάλεια στην αγορά. Βλέπουμε λοιπόν Ε, πως ε, και μέσα σε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως οι εξαποστάσεως ε, πωλήσει αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία και της δίνεται και η απαραίτητη έμφαση μέσα σε αυτή την πρόταση. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επικοινία, η ο πολυδιάστατο χαρακτήρα τη εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάντα μιλάμε για το γνωστικότητα και ούτω καθεξή, αλλά θα πρέπει να ληφθεί και αυτή η υπόψη και να ενδυναμωθεί αλλά το ερώτημα βέβαια είναι το κατά πόσο η Ευρώπη είναι σήμερα αρκετά όρημη για μια τέτοια πρόταση. Εάν δηλαδή ε, τα δικαιώματα που προβλέπονται στην νομοθεσία ε, θα συνοδευτούν από μια αντίστοιχη εφαρμογή ε, αυτής της νομοθεσίας με βάση και βέβαια την εθνική νομοθετική παράδοση και με βάση τα δικαιώματα προστασίας του κανονικού που προβλέπονται. Νομίζω πως ένας κώδικας λοιπόν του δικαιωμάτου του καταναλωτή θα πρέπει να ε, προσανατολίζεται ε, σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι στα συμφέροντα των 27 διαφορετικών ε, κρατών μελών. Να μην έχουμε ένα melting pot δηλαδή όπως λένε οι Αμερικάνοι, αλλά να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, ένα σύστημα το οποίο πραγματικά θα βρίσκεται κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, έχουμε δηλαδή μακροπρόθεσμους στόχους οι οποίοι σχετίζονται με την παρούσα πρόταση, αλλά είναι και λίγο αντιφατική κάποιες ε, φορές ε, με αυτήν. Ε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της νομοθετικής αναρμόνισης και το τι επιτυγχάνεται εκεί. Το ερώτημα δηλαδή που τίθεται για μας είναι το τι μπορούμε να επιτύχουμε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια με αυτή την πρόταση και από την πλευρά μας μα Επιτροπή. Εμεί θα προσπαθήσουμε να συμμετάσχουμε επικοδομητικά σε όλη αυτή τη συζήτηση και Χαίρομαι το γεγονό ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν με αυτήν την ε, ακρόαση τη δυνατότητα να συζητήσουν εκ νέου όλα τα υπέρ και τα κατά αυτή τη ε, νέα ε, πρόταση και θα ήθελα να σα προτείνω, αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, με βάση τα όσα συζητηθούν και σήμερα μέχρι ε, μέσα η τέλη Νοεμβρίου να συνταχθεί ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική μας προσέγγιση για αυτό το ζήτημα. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που είχα δυνατότητα να πάρω το λόγο για αυτό το ζήτημα σήμερα. Αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση και βέβαια τα... αναμένω πως θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. για την ε, ισχυρή καθοδηγητική σου στάση όσον αφορά το θέμα αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με την πρώτη παρουσίαση. Ο τρόπο με τον οποίο διαθρώσαμε την ε, ακρόαση σήμερα έχει ω εξή. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε παρουσίαση τη Επιτροπή δίνοντα ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα συμπληρωματικά έγγραφα που πήραμε και στα ε, ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Μετά θα έχουμε ένα σύντομο διάστημα ερωτήσεων και στη συνέχεια ζητήσαμε από τον καθηγητή Σούλτεν και από το Πανεπιστήμιο του Όσναμπρουκ να μας μιλήσει για τα νομικά πλαίσια και να μας κάνει μια διορθωτική ανάλυση για 10 λεπτά και στη συνέχεια θα έχουμε ερωτήσει. Μετά έχουμε μια ε, τέσσερα άποψη των καταναλωτών και των επιχειρησεων ερωτήσει ερωτήσεις-απαντήσεις και τέλος ε, το καταληκτικό τμήμα από τον Άντερ το οποίο θέλω να τον καλωσορίσω θερμά, ο σύμβουλο για θέματα καταναλωτών ε, της, ε, από την σφιντική κυβέρνηση εδώ στις Βρυξέλλες, ο παρακολουθεί το θέμα με πολύ μεγάλη προθυμία. Φαίνεται ότι ε, ε, έρχεται στην Επιτροπή μας σχεδόν όσο συχνά όσο και εγώ. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορά. Και τώρα να προχωρήσουμε με τις εργασίες μας. Κυρία Τεστόρη Κότζη, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω εδώ για άλλη μια φορά και θα σας δώσω το λόγο για να μας μιλήσετε για την πρόταση και για το νέο υλικό το οποίο μας στείλατε σήμερα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Σιγητά και μέλη του Κοινοβουλίου. Εμείς ε, σίγουρα χαιρόμαστε ιδιαίτερα με την ακρόαση αυτή. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή και εξελογούμε αυτή την ευκαιρία για να σας εξηγήσουμε περαιτέρω την πρότασή μας και ταυτόχρονα θέλουμε να ακούσουμε τι δικέ σα θέσει των διαφορών μελών του Κοινοβουλίου και των όλων των ενδιαφερομένων. Για μα αυτή η πρόταση είναι μια βασική πρωτοβουλία. Για τον Επίτροπό μου είναι βασική πρωτοβουλία γιατί πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη οδηγία όταν θα εγκριθεί θα ε, αποτελέσει σημαντική συμβολή προς την ιστορική αγορά. Θα αυξηθεί ο ανταγωνισμό, ο ανταγωνισμός και θα οδηγήσει σε καλύτερες τιμές και σε περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές. Όπως είπε και ο εισηγητής, σαφώς πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις νόμιμες προσδοκίες και τις θεμητές προσδοκίες των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Μόνο η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών και νομική, αβεβαιότητα, νομική βεβαιότητα που θα προκύψει από την πλήρη εναρμόνιση, μόνο λοιπόν με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους δύο στόχους που μόλις ανέφερα. Επιτρέψτε μου να κάνω μια μεταφορική ε, ε, μια μεταφορά. Ε, θα έχουμε, με την πρόταση αυτή θα έχουμε μια, ένα νησί βεβαιότητας μέσα σε ένα ωκεανό αποκλίνουσών εθνικών νομοθεσιών. Όπως είπατε λοιπόν και εμείς πιστεύουμε ότι η ιστορική αγορά πρέπει, αξίζει να ξεκινήσουμε και αξίζει να ξεκινήσουμε με αυτό το μικρό νησί. Θα και ε, η Επιτροπή θα δείξει ευελιξία και όσον αφορά το περιεχόμενο τη πρόταση, αλλά και όσον αφορά το επίπεδο προστασία. Δηλαδή, θέλουμε ώστε να δουν υψηλότερο επίπεδο. Αλλά ε, ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο βασικό μα στόχο είναι να ε, απομακρύνουμε τον κατακαιρματισμό σε νομικό επίπεδο των κανόνων προστασία του καταναλωτή, που κατά την άποψή μα αποτελεί αυτό ο κατακαιρματισμό εμπόδιο σωστή λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι έτοιμη να δεχθεί ε, οτιδήποτε λιγότερο από ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα ισχύει για όλους τους καταναλωτές και για όλους τους επιχειρηματίες. Κοιτάξτε, ακούμε επικρίσεις από τότε που να επιτάπητο στην πρόταση αυτή. Και ε, ε, γνωρίζουμε ότι πολλοί, αλλά ε, γνωρίζουμε ότι πολλοί υποστηρίζουν. Αυτό μου δεν σημαίνει ότι την πρότασή μας, ότι όλοι έχουν καταλάβει τις πιθανές, τα πιθανά οικονομικά ωφέλη που θα προκύψουν. Γιατί κατά την αξιολόγηση αντικτύπου κάναμε μία σε βάθος ανάλυση της οικονομικής των οικονομικών επιπτώσεων της πρότασης, βεβαίως με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία δεν ήταν οριστικά και πλήρη. Όπου υπάρχουν τομείς που παρουσιάστηκε ανεπαρκή σε πληροφόρηση, ε, εκεί θέλουμε να διευρύνουμε τις γνώσεις μας. Και στο τέλος του χρόνου θα παρουσιάσουμε μια μία μελέτη για ένα τομέα στον οποίο έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν ελλείψεις, που αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιδρούν Ε, ε, και, το πώς βλέπουν δηλαδή ε, τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους στην περίπτωση των ελαττωματικών αγαθών. Δηλαδή, τι προτιμά ο καταναλωτή με δύο λόγια. Επιδιόρθωση, ακύρωση τη σύμβαση, επιστροφή. Εδώ λοιπόν δεν γνωρίζουμε ακόμα απόλυτα ποια είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών. Και αν το ΜΠΕΚ και οι άλλε οργανώσει των καταναλωτών έχουν συγκεκριμένε απόψει, ε, καταλαβαίνετε ότι είναι ευπρόσδεκτε. Μας ζητήθηκε η, ε, η μελέτη ε, της ε, πρότασης αυτής επί των εθνικών νομοθεσιών. Γι' αυτό σας στείλαμε το συγκριτικό πίνακα. Κοιτάξτε, η εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Μην αρχίσετε να μετράτε τα συν και τα πλήν, γιατί το αποτέλεσμα δεν θα οδηγήσει πουθενά. Σας το ξαναλέω, δεν είναι ε, το οριστικό αποτέλεσμα. Και είμαστε ανοιχτοί και στα κράτη-μέλη και στι οργανώσει των επιχειρήσεων και στι οργανώσει των καταναλωτών και θέλουμε να μα βοηθήσετε να συμπληρώσουμε αυτό το συγκριτικό πίνακα. Γιατί αν θέλουμε να καταλάβουμε το πραγματικό αντίκτυπο αυτή τη οδηγία σε εθνικέ νομοθεσίε, τότε πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση. Δεν θέλουμε λοιπόν η συζήτηση να συγκεντρωθεί στο έγγραφο αυτό, αλλά στην ίδια την πρόταση. Όσον αφορά την πρόταση, να σας πω ότι τρει είναι οι βασικοί τομεί ανησυχίας για μας και φαντάζομαι και για εσάς. Πρώτα απ' όλα, το πεδίο εφαρμογή. Εμείς πιστεύουμε σαφώς ότι η συσχέτιση ανάμεσα στην πρόταση αυτή και ε, το παραδοσιακό εθνικό ενοχικό δίκαιο πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω και θα συνεργαστούμε μαζί σας και με το Συμβούλιο για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ιδιαίτερα σε σχέση με ε, την, ε, ε, με την αποζημίωση σε περίπτωση ελαττωματικών αγαθών. Το ξαναλέω. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε μία διάταξη στην πρόταση, όπου επιβεβαιώνουμε σαφώς ότι η πλήρης εναρμόνιση ε, των δράσεων αυτών αποκατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικών αγαθών δεν, γίνεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας ε, του ενοχικού δικαίου, του δικαίου περισυμβάσεων. Στη συνέχεια να σας πω ότι η Επίτροπός μου, η Επίτροπος Κούνεβα, είναι έτοιμη, έτοιμη να προχωρήσει περισσότερο προς την κατεύθυνση ε, της ε, περαιτέρω ρύθμισης για τα ελαττωματικά αγαθά και της διεύρυνσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Στο Συμβούλιο, ε, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τα θέματα αυτά, γίνονται συζητήσεις, διερευνητικές συζητήσεις, για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε στην ίδια την πρόταση δικαίωμα απόρριψης, επιστροφής, όπως, ε, όπως συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ε, δικαίωμα ε, παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Τώρα, τρίτο σημείο. Σαφώ η πλήρη εναρμόνιση θα έχει επιπτώσει στου εθνικού κανόνε που αφορούν την, τους αθέμιτους συμβατικούς όρους. Και εδώ να σας πω ότι τα κράτη-μέλη, αν εγκριθεί η οδηγία, θα πρέπει να τροποποιήσουν ε, τον υφιστάμενό τους ε, ε, κατάλογο όσον αφορά τις αφέμητες, τους αφέμητους συμβατικούς όρους. Είναι σαφές. Πρέπει να, με βάση τη νέα νομοθεσία, θα αλλάξουν τους καταλόγους στα τα κράτη-μέλη. Όμως η πρόταση δεν θα θέσει αμφισβήτηση την υφιστάμενη εθνική νομολογία για τους αθέμητους όρους και κυρίως δεν πρόκειται να περιορίσει την αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να ε, διερευνούν ε, τους ε, όρους της σύμβασης. Η γενική λοιπόν ρήτρα θα έχει αυτόνομη ρυθμιστική λειτουργία. Όπως σας είπα, αυτά για μας τα τρία ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογής. Δεύτερον, η σχέση με το παραδοσιακό εθνικό ενοχικό δίκαιο. Και τρίτον, οι εθνικοί κανόνες των αθέμητων συμβατικών όρων. Τώρα, σας λέω ότι ε, αυτά είχα να πω αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Περιμένουμε με ανυπομονησία τη συζήτηση και είμαστε σίγουροι ότι σε αυτή την νομοθετική διαδικασία με το Κοινοβούλιο και με τη συγκεκριμένη επιτροπή σας θα βελτιώσουμε την πρότασή μας. Ευχαριστώ. thank you very much indeed. Ευχαριστούμε πολύ για τη σαφέστατη περιγραφή σας. Σημείωσα την ε, πολύ ωραία σας περιγραφή για ένα νησί βεβαιότητα σε μια θάλασσα αβεβαιότητας. Το ερώτημα βεβαίως είναι πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι αυτή η νησίδα και πόσο πολύ νερό θα το περικυκλώνει. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ο κύριος η εισηγητής, ε, θα θέλει σίγουρα να θέσει ερωτήσεις. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Σφάμπ, μετά στον κύριο Τριανταφυλλίδη και μετά σε όποιον άλλον θέλει το λόγο. Θα περιμένω λίγο πριν κλείσω την λίστα. Αλλά θα ακούσουμε πρώτα όλες τις ερωτήσεις και μετά θα απαντήσει η κυρία Τεστόρη. Άντρες, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πολύ σαφή περιγραφή της Επιτροπής. Δύο ερωτήσεις η πρώτη μας επιστρέφει στο σημείο εκκίνησης, ε, δηλαδή το κατά πόσο είναι σαφές το πεδίο εφαρμογής. Υπάρχουν ε, σαφείς ενδείξεις ότι η εθνική νομοθεσία για τις ε, συμβάσεις των καταναλωτών θα παραμείνει αναλύωτη. Άρα δεν πρόκειται να έχουμε την ε, ολοκλήρωση της αγοράς που Επίση, ασχέτως μεγέθους, να μπορούν να διοχετεύσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι όμως αυτός ο στόχος εφικτός με την προτινόμενη οδηγία. Καταρχήν, θα πρέπει να εξετάσουμε το επίπεδο εναρμόνισης. Η πρόταση ορίζει την αρχή της πλήρους εναρμόνισης, δηλαδή της εφαρμογής κανόνων που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς τη δυνατότητα εξαίρεσης. Μέσα από την πλήρη εναρμόνιση επιδιώκεται ουσιαστικά η εφαρμογή κατώτατων ορίων σε τομείς όπως οι εγγυήσει προϊόντων για να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο στα προϊόντα τους ανεξαρτήτως σε ποια χώρα τα πολλούν. Με αυτή τη ρύθμιση η προστασία των καταναλωτών στις πλήστες χώρες τίθεται σε κίνδυνο αφού τα δύο χρόνια περίοδος εγγύησης αποτελούν πλέον την οροφή για όλα τα προϊόντα και συνεπώς σε πολλούς τομείς μειώνουν την περίοδο εγγύησης για τους καταναλωτές. Υπάρχει πληθώρα προϊόντων, παραδείγματο χάρη ηλεκτρικές συσκευές, που συνοδεύονται επί του παρόντος με μακρότερη περίοδο εγγύησης. Δημιουργούνται με αυτή τη ρύθμιση οι προϋποθέσεις εμπορίας συμβάσεων εγγύησης μεγαλύτερης των δύο ετών. Συνεπώς μια εταιρεία που πολλούσε μια ηλεκτρική συσκευή με πέντε χρόνια εγγύηση θα έχει την δυνατότητα να απολύει τη συσκευή με δύο χρόνια εγγύηση και να διαθέτει επιπλέον προς πώληση τη δυνατότητα αναβάθμισης της εγγύησης στα πέντε χρόνια. Άρα μέχρι τώρα η υποχρέωση του κατασκευαστή αποτελεί πλέον προϊόν της πώληση. Σε άλλε διατάξει, σε περίοδο υπαναχώρησης για τι εξαποστάσεω συμβάσει και τι συμβάσει εκτό καταστήματο, αποτελεί. Συγγνώμη, αλλά έχουμε ακρόαση και θέλουμε να ακούσουμε ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Είναι ενδιαφέρον η δήλωσή σας, αλλά υποθέτω ότι έχετε να κάνετε και κάποιες ερωτήσεις. αποτελεί κεφαλαιόδες ζήτημα. Δεν είμαστε αρνητικοί στις προσπάθειες βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου. Ε, αντίθετα το επιδιώκουμε, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται με προστασία των καταναλωτών και όχι των επιχειρήσεων. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διάθεση να ακούσει του συνδέσμους καταναλωτών και να προχωρήσει σε ρύθμιση με βάση τι δικέ του ανάγκε ή θα γίνει και πάλι η αιτία να ενισχυθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να δεσμεύουν του καταναλωτέ με δυσμενέστερου όρου. Γιατί δεν υπάρχει πρόταση από πλευρά Επιτροπή που να οθεί την μείωση των τιμών των αγαθών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την ερώτηση. Ευχαριστώ. Όλοι θέλουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, εγώ προσωπικά δεν βλέπω ποια είναι τα ουσιαστικά κέρδη για τους καταναλωτές της Ευρώπης. από δανεική πρόπτικη για παράδειγμα. Ποιο είναι το κέρδος για τον καταναλωτή. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, συγκριτική ανάλυση. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε επίσης να πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα μέσα στο σχέδιο πρότασης που δεν βρίσκω απόλυτα σωστά. Ειδικά όσον αφορά τις συγκρίσεις μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής αρμοδιότητας, και σίγουρα αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι οι επικαλύψεις. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει ανοιχτός διάλογος έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Um, θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Τεστόρη να απαντήσει σε αυτά τα τρία ερωτήματα, αλλά έχουν επίσης ζητήσει το λόγο οι κύριοι Λάιγναρ και Βάιλερ. Α, έχουμε επίσης RL, οπότε αυτοί θα πάνε σε ένα δεύτερο γύρο. Μπορείτε να απαντήσετε κυρία Τεστόρη. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω μια γενική απάντηση και μετά θα ζητήσω από το συνάδελφο που ασχολείται με θέματα εθνικών κρατών να απαντήσει στις περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούσαν κυρίως τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, δεν θα έχουμε πλήρη εναρμόνιση. Αυτό αποτελεί ένα ουσιώδες σημείο της πρότασης, αλλά δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να επικρίνουμε την πρόταση. Ακόμη και αν κατορθώσουμε να εναρμονίσουμε μόνο ορισμένα τμήματα των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, πάλι δημιουργείται νομική ασφάλεια που θα ενισχύσει το ενδοκινοτικό εμπόριο. Σε κατάσταση οικονομικής κρίσης χρειαζόμαστε μια πιο αποτελεσματική εσωτερική αγορά. Μέσω λοιπόν αυτής της νομικής ασφάλειας για τις επιχειρήσεις θα μπορέσουμε να απελευθερέσουμε επιπλέον την αγορά, να ανοίξουμε την αγορά, κάτι που τελικά θα είναι καλύτερο για τους καταναλωτές. Και μετά θα δώσω το λόγο και στο συνάδελφο για να σας μιλήσει ακριβώς για τη σχέση εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το άλλο ερώτημα είναι αν θέλουμε πλήρη εναρμόνιση ή όχι. Όταν η Επίτροπος κατέθεσε την πρόταση, ήθελε πλήρη εναρμόνιση. Για τους λόγους που είπα και πριν. Γιατί θα έχαμε τελικά μία ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά χωρίς σύνορα όπως ισχύει σήμερα και χωρίς περιορισμούς. Τώρα, γιατί χρησιμοποίησαμε επιτροπολογία, γκρίζα λίστα, μαύρη λίστα. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή όπου πάντα τα νομοθετικά όργανα θέλουν να έχουν πολλές αρμοδιότητες. Γιατί ξεκινάμε από διάφορες γνωστές δεδομένες πρακτικές. Εδώ όμως θέλουμε να μπορούμε να τροποποιούμε συχνά και αυτό μέσω διαδικασίας συναπόφασης είναι σχεδόν αδύνατο. Επαναλαμβάνω όμως, τον πίνακα μην τον χρησιμοποιήσετε ως βάση για να μετρήσετε ποια θα είναι τα ουσιαστικά ωφέλη, γιατί χρειάζεται συμπλήρωση. Χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Τζουζέπε Βεμόντε, ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να σας απαντήσει στα πιο νομικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω συμπληρώνοντας τα όσα είπε η κυρία Τεστόρη στην απάντηση προς τον εισηγητή ποια είναι η σχέση της οδηγίας με την ε, γενική συμβατική νομοθεσία των κρατών μελών. Και ποιο είναι το, έφε, το όφελος που θα έχουμε αν δεν αλλάξουμε την νομοθεσία των κρατών μελών. Κάτι που πρέπει να προσέξετε και το οποίο έχουμε προσέξει πολύ είναι η σχέση με τα ένδικα μέσα για την συμβατική νομοθεσία, για παράδειγμα για τα ελαττωματικά αγαθά. Προσπαθούμε να δούμε ποια θα είναι η διασύνδεση με τις γενικές ρήτρε όσον αφορά τη συμβατική νομοθεσία. Να πω ότι σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν δύο επίπεδα για ένδικα μέσα. Τα γενικά μέσα για μέσω της συμβατικής νομοθεσίας και αυτά που αφορούν τους καταναλωτές που είναι πιο επωφελή για τους καταναλωτές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με αυτή την οδηγία είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση για τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές χωρίς να αλλάξουμε τα γενικά. Και θέλουμε να έχουμε μία εξελιτική εναρμόνιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών όταν έχουν ένα ελαττωματικό προϊόν στα χέρια τους. Αν μας δώσει αυτή τη δυνατότητα το Συμβούλιο, τότε θα προσθέσουμε και άλλα δικαιώματα για τους καταναλωτές στην πρόταση, έτσι ώστε να εναρμονίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα μέσα προσφυγής του καταναλωτή σε περίπτωση που αγοράσει ελαττωματικό προϊόν. Το άλλο που ανέφερε ο εισηγητής ήταν η σχέση μεταξύ μαύρης και γκρίζας λίστας καθώς και με την ε, ρήτρα περί αθέμητων πρακτικών. Καθώς επίσης και το τι μας προσφέρει εδώ η Επιτροπολογία. Η προστιθέμενη αξία της επιτροπολογίας είναι να μας επιτρέπει στο μέλλον να αντιμετωπίζουμε άμεσα αναδιόμενες αθέμητες πρακτικές, αναδιόμενες νέες αθέμητες συμβατικές ρήτρες. Να μπορούμε άμεσα να τις προσθέτουμε στη μαύρη και την γκρίζα λίστα. Να πω εδώ ότι η μαύρη και η γκρίζα λίστα δεν είναι εξαντλητικοί κατάλογοι, δεν αναφέρουν όλα τα κείμενα, τα πιθανά περιέχουν αθέμητες ρήτρε. Απλά είναι ένα δίκτυο, ένα δίκτυ ασφαλείας και βεβαίως ακόμη και αν μια πρακτική δεν αναφέρεται στη μαύρη την κρίζα λίστα, παρόλα αυτά μπορεί αυτή η ρήτρα να συμπεριληφθεί στις αθέμητες πρακτικές με βάση το γενικότερο κείμενο, τη γενική ρήτρα. Έχουμε λοιπόν και τη γενική ρήτρα για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και την μαύρη και την κρίζα λίστα που λειτουργούν συμπληρωματικά. Τώρα, ποιες θα είναι οι συνέπειες της οδηγίας στις εμπορικές πρακτικές. Να πω ότι η οδηγία απευθύνεται στα κράτη-μέλη, άρα δεν εμποδίζει μεμονωμένες επιχειρήσεις να προχωρήσουν παραπέρα και να δώσουν και άλλα δικαιώματα στους καταναλωτές. Ίσα ίσα που ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Τέλος, όσον αφορά το όφελος για τους καταναλωτές, πέρα από τον πίνακα, ας θυμόμαστε ότι ο κανονισμός Ρώμη 1 θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους και εξαιτίας του θα ζητείτε συμμόρφωση με τις νομοθεσίες 27 κρατών μελών. Αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στους καταναλωτές, αυτός ο κατακαιρματισμός, αν δεν κάνουμε κάτι για να αντιδράσουμε. Σας ευχαριστώ. Όπως σας είπα, έχουμε τρεις ακόμα ερωτήσεις. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι και συγκεκριμένοι. Κύριε Λέχνερ, κυρία Βάιλερ και κύριος Άριος. Πρώτα ο κύριος Λέχνερ. Ε, ε, ganz kurz, es ist äh, gerade eben er Πολύ σύντομα. Ε, έγινε μια αναφορά στο Εθνικό Ενωσικό Δίκαιο και αυτό με βρίσκει αλλά θα σύμφωνο, αλλά θα ήθελα να ακούσω κάποια παρατήρηση ω ε, προ ε, το πώ φαντάζεσαι όλε αυτέ τι ε, εργασίε στο γενικότερο πλαίσιο του CFR. Και α, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Η κυρία Τεσόρη είπε κάτι σε σχέση με, τις, με τους αθέμετους όρους στα συμβόλαια, ότι αυτό δηλαδή μπορεί να εναρμονιστεί πλήρω σε αυτό το τομέα. Αλλά αν έχουμε μια τέτοια ολοκληρωμένη εναρμόνιση, τότε φοβούμε ότι ενδεχομένω να φτάσουμε στην κατάσταση όπου κάθε μεμονωμένη περίπτωση να καταλήγει στο δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δηλαδή, τι ακριβώ θα συμφίσει σε αυτή την περίπτωση, ή ενδεχομένω έχω κάνει κάποια παρανόηση. Εν πάση περιπτώσει, πού βρίσκονται τα εθνικά περιθώρια και πού θα καταλήγουν τέτοιου είδου υποθέσει τελικά. Ευχαριστώ. Κυρία Βάιλα, έχετε λόγο. Ναι, και στη δική μου προσοχή υπέπεσε αυτό ότι ε, πριν από τι εκλογές είχαμε συζητήσει ε, και ε, την νομοθεσία σε ό,τι αφορά τι αθέμητε εμπορικέ ε, πρακτικέ και το κατά πόσο αυτή εφαρμόζεται ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η σχέση τη ε, με αυτήν την ε, νέα πρόταση, της, αυτή τη νέα οδηγία. Δηλαδή, άλλοι επικαλύπτονται, είναι αλληλοσυμπληρωματικέ. Ήδη ρωτήθηκε τέτοια το ερώτημα του κατά πόσο είναι λίγο πρόωρη αυτή η φάση για μια πλήρη εναρμόνιση ε, επιτρέψτε μου εγώ να κάνω και μια προσθήκη. Ίσως πράγματι η εναρμόνιση να είναι ε, μια ενδιαφέρουσα προοπτική ε, για όλους, αλλά ίσως δεν έχει οριμάσει επαρκώς εν λόγω πρόταση οδηγίας, γιατί και από τη δική σας πλευρά, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν τονίζονται ιδιαίτερα ή δεν διαγράφονται ιδιαίτερα τα πλέον εκτήματα. Ε, ήδη έχουμε συζητήσει επανειλημμένα ότι χρειάστηκε να προωθήσετε ενεργά τη δική σα πρόταση, να την διαφημίσετε εντό εισαγωγικών, όχι τόσο σε εμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και σε άλλου φορεί, τη μη κυβερνητικέ οργανώσει και ούτω καθεξή. Πράγματι έχουμε κάποιο οικονομικό όφελο, αλλά αυτό δεν επαρκεί από μόνο του. Θα ήθελα δηλαδή να έχουμε και κάποια επιπρόσθετη χρησιμότητα, κάποια ευρωπαϊκή υπεραξία για κάτι τέτοιο και όχι απλά μερικά σέντα, οποία θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε. Και δεν επαρκεί το να λέμε ότι θα υπάρξει μια προσέγγιση μεταξύ του επίπεδου της Δανίας και του επίπεδου ε, της Λιθουανίας, στο προτύπο εκεί. Αυτό είναι ε, θετικό μεν, είναι θετικό να ακολουθούμε αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό χρειάζεται ίσως 20 χρόνια να συμβεί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι απλά. Τι σα έχει το λόγο. Τελευταία ερώτηση, ο κύριο Άρη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, με βάση όλα αυτά που άκουσα σήμερα για τα δικαιώματα του καταναλωτή, να σα πω το εξή. Δεν άκουσα τίποτα για τους καταναλωτές στο διαδίκτυο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσον αυτή η οδηγία θα λάβει υπόψη της και το ζήτημα αυτό και θα προβεί προς κάποια ρύθμιση προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί η άποψή μου είναι ότι εδώ έχουμε μια αγορά με πολλές δυνατότητες στην Ευρώπη και θα πρέπει τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί ε, να έχουν τις ίδιες ε, ε, εγγυήσεις από νομική άποψη με τους παραδοσιακούς καταναλωτές. Με αυτή την έννοια υποβάλλω μια πρόταση στην Επιτροπή να προταθεί ε, μια εμπορική εγγύηση, σφραγίδα εμπορικής εγγύησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ε, τις νομικές εγγύησεις που θα έχει και ο καταναλωτής που ε, αγοράζει μέσω του διαδικτύου. Ευχαριστώ. Well, thank you uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τεστόρη, ξεκινήστε και ίσως συνεχίσει ο συναδελφός σας. Σα ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στην πρώτη ομιλήτρια, στη δεύτερη μάλλον ομιλήτρια, σχέση με, τα, με τις ανησυχίες των καταναλωτών. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι θεμητές ανησυχίες του καταναλωτή όσον αφορά ορισμένες ε, διατάξεις οδηγίας. Και όπως είπα, ε, η Επιτροπός μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή στη συζήτηση. Όλοι μας ε, θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματα που υπάρχουν ιδιαίτερα όσον αφορά δύο από τις διατάξεις αυτές, για να υπάρξει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας το χρονικό διάστημα ισχύω εγγύηση και τα ένδικα μέσα. Θα τα μελετήσουμε αυτά τα ζητήματα για να καταλάβουμε και τι απόψει των καταναλωτών. Πιστεύω λοιπόν ότι Μπορώ να σα πω το εξή. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να διευκρινιστούν και ορισμένα πράγματα στα οποία και εμείς θα θέλαμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Και θέλουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί σας για να μπορέσουμε να επιφέρουμε τις κατάλληλες βελτιώσεις. Όσον αφορά το περιθώριο εγκληγμών για τα κράτη-μέλη και η σύνδεση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο Τζουζέπε θα απαντήσει. Ευχαριστώ, Πάολα. Ξεκινούμε με την τελευταία ερώτηση. Κοιτάξτε, μεγάλο μέρος της πρότασης αφορά τις συμβάσεις εξ που συμπεριλαμβάνουν και τις συμβάσεις μέσω του διαδικτύου. Όλες λοιπόν οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του διαδικτύου, όλες οι αγορές που γίνονται μέσω του διαδικτύου υπόκειται στις διατάξεις οδηγίας. Ο καταναλωτής όταν αγοράζει κάτι εξ που καλύπτει και την περίπτωση αγορών μέσω του διαδικτύου, ε, ε, χέρι περαιτέρω προστασίας σε σχέση με την παραδοσιακή αγορά στο κατάστημα. Δηλαδή, ε, εδώ οι απαιτήσει για πληροφόρηση είναι πιο αυστηρές, έχει και το, και το δικαίωμα υπαναχώρησης ε, μέσα σε 14 ημέρες αν δεν του αρέσει το προϊόν, χωρίς να δικαιολογήσει καθόλου την, το, το, το, το, ότι άλλαξε άποψη. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Λέχνερ, ε, σε σχέση με το κοινό πλαίσιο αναφοράς, προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε αυτά τα δύο σχέδια που είναι δίδυμα. Το κοινό πλαίσιο αναφοράς και ένα αναθεώρηση του εκτιμένου. Ε, ε, πρέπει να σας πω ότι ήμουν πρόεδρος σε μία σειρά από εργαστήρια των εμπειρογνωμόνων στο κοινό πλαίσιο αναφοράς και τα ευρήματα ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση της οδηγίας. Άρα έχουν ληφθεί υπόψη. Η πρόταση βέβαια δεν σέβεται πάντα ή δεν αντικατοπτρίζει πάντα τα ευρήματα αυτών των, ε, ε, των εμπειρογνωμόνων. Τώρα έχουμε ε, το ακαδημαϊκό κοινό πρόγραμμα πλαίσιο αναφορά και θα φροντίσουμε έτσι ώστε η τελική εκδοχή της οδηγίας να είναι συνεπής με την τελική εκδοχή του κοινού ε, πλαίσιο αναφορά. Θα υπάρξει λοιπόν απαραίτητα ε, συσχέτιση και στοιχεία των δύο σχεδίων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι στο τέλο ε, υπάρχει ε, εξασφαλίζει η συνολική συνοχή. Τώρα, ορισμένα ζητήματα είναι εθνικά. Αυτό που είπατε δηλαδή για την προσθέμενη αξία, για την πλήρη εναρμόνιση. Μα κοιτάξτε, δεν πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό κώδικα. Ο εθνικό νομοθέτης είναι αυτό που θα φροντίζει έτσι ώστε οι πλήρω εναρμονισμένε διατάξει οδηγία εντάσσονται στα γενικά πλαίσια του αστικού δικαίου της χώρας. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Ε, υποχρεώσεις των μερών όταν αποσύρεται από τη σύμβαση, η παραχωρία από τη σύμβαση ο καταναλωτής. Δεν λέμε όμως τι γίνεται σε περίπτωση που δεν επιστρέφει έγκαιρα στον έμπορο καταναλωτής. Και δεν λέμε επίσης τι θα συμβεί αν ο έμπορος δεν επιστρέψει τα χρήματα τα οποία κατέβαλε ο καταναλωτής. Αναπόφευκτα όλα αυτά τα ζητήματα. Διαφορετικά θα ήταν 100 ε, φορές ε, πιο μακροσκελής η οδηγία. Αυτά τα ζητήματα ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τις ζημιές, λέμε ότι αν υπέστη ζημία ο καταναλωτής λόγω του ε, ελαττωματικού αγαθού, το κράτος μέλος θα ρυθμίσει το δικαίωμα αποζημίωσης για τις ζημιές. Αλλά όλοι αυτοί οι όροι και τα λοιπά, οι προϋποθέσεις θα ρυθμίζονται από τον εθνικό νομοθέτη. Και ακριβώ γι' αυτό ακολουθήσαμε την οδό τη οδηγία και όχι του κανονισμού. Γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο για τον εθνικό νομοθέτη να τα συμπεριλάβει όλα αυτά ε, στον αστικό κώδικα. το, τη σχέση τώρα με την ε, οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και αυτό που είπε η κυρία Βάιλερ. Προσπαθήσαμε να το απαντήσουμε στο συνοδευτικό σημείωμα, στο σημείωμα που συνόδευσε τον στο συγκριτικό πίνακα. Ε, η, η οδηγία αυτή ε, δεν είναι οδηγία που αφορά τον αρχικό δίκαιο, αλλά την αγορά. Ο καταναλωτής δηλαδή υπό την ιδιότητά του του αποδέκτη ε, της εμπορικής πρακτικής. Και όχι, η οδηγία δεν ε, ε, προστατεύει τον επιμέρους καταναλωτή αν θέλετε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να λάβουμε υπόψη την οδηγία για τις αφέμιτες εμπορικές πρακτικές που δεν εκχωρεί ε, επιμέρους δικαιώματα στους καταναλωτές. Σε αυτή την πρόταση λοιπόν έχουμε ορισμένε απαιτήσει και ε, και ε, ε, έχουμε δώσει μέσα απαιτήσει ε, για, για τις πωλήσει που ταυτίζονται σε κάποιο βαθμό με, τις, με ορισμένα πράγματα που αναφέρει η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Παράδειγμα, όταν ε, έχουμε αθέμητες πρακτικές στην περίπτωση που απευθύνεται στον αγοραστή ο πολιτής, ε, τότε εκεί τα πράγματα είναι κοινά. Δηλαδή προστατεύουμε και τα συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών που κάνει η άλλη οδηγία, αλλά και τα επιμέρους συμφέρον των, των καταναλωτών με τη συγκεκριμένη οδηγία. Ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω πως θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε πιο γενικά ερωτήματα ε, στο μέλλον. Να σας ευχαριστούμε ε, και για τις παρεμβάσεις σας και για τα εγγραφά σας τα οποία νομίζω έχουν διανεμηθεί και είναι στη διάθεση όλων εδώ. Ε, βρίσκονται στο public domain τους άλλους για να μπορέσετε να τα εξετάσετε. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο στοιχείο το προσεζήτηση με τον τίτλο «Δομική ανάλυση του νομικού πλαισίου» «Structural Analysis of the Legal Context» ε, πράγμα βέβαια το οποίο σχετίζεται και με την ε, σχέση μεταξύ του κοινοτικού δικαίου του εναρμονισμένου, ε, της εναρμονισμένης νομοθεσίας και της νομοθεσίας των κρατών και ελπίζω πως ο καθηγητής ε, Δ. Hans Σούλτεν Nolke ε, θα μπορέσει να μας ε, βοηθήσει με μια παρέμβαση για να βρούμε εδώ, να, βγάλουμε κάποια άξιση σχέση με αυτό το ζήτημα και μάλιστα μόνο μέσα σε 10 λεπτά θα πρέπει να το κάνει για να έχουμε και στη συνέχεια κάποιο χρόνο για συζήτηση. Έχετε το λόγο λοιπόν κύριε Σωτέ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε, ελπίζω να τα καταφέρω. Όπως γνωρίζετε, εξωτιμητήρες και κύριοι, η πρόταση αυτής της ε, οδηγίας ε, εκλήθηκε με πολύ επιφύλαξη από τον ε, νομικό κλάδο. Σχεδόν κανείς δεν έχει ταχθεί υπέρ αυτής της πρότασης και κάποιες φορές ήταν καταστροφική η κριτική η οποία στήθηκε. Τρίαντα κυρία σήμερα. Καταρχήν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα νομοτεχνικά αν θέλετε τα οποία είναι ιδιαίτερα προβληματικά και από εκεί και μετά το μεγαλύτερο ακόμα πρόβλημα η οδηγία ε, έχει πολύ αρνητικές, ίσως και καταστροφικές ε, συνέπειες ε, σε έναν ευρύτερο τομέα και σε ένα ευρύτερο πεδίο και όχι μόνο σε αυτό στο οποίο περιορίζεται. Ενώ τίθεται και το ερώτημα του κατά πόσο θα παραμένει το επίπεδο προστασία στο καταναλωτή εκεί που βρίσκεται σήμερα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εγώ να πω ευθύ εξ αρχή ότι η δική μου στάση δεν είναι τόσο επικριτική. Θεωρώ δηλαδή πως ε, μπορεί να σωθεί αυτή η πρόταση και ενδεχομένως μπορούμε να επιτύχουμε ε, κάτι από εδώ και από εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της. Είναι πολύ σημαντικό ε, να πούμε με σαφήνεια το γιατί καταρχήν χρειαζόμαστε μια τέτοια οδηγία. Να εξετάσαμε λοιπόν τις τέσσερις οδηγίες οι οποίες γίνεται η προσπάθεια να συγχωνευτούν και να ενσωματωθούν κατά κάποιο τρόπο σε μια και είδαμε ότι πράγματι είναι τόσο πολυδιάστατη εικόνα στα διάφορα 27 κράτη-μέλη έτσι ώστε να είναι πραγματικά αδύνατο ουσιαστικά να μπορεί κανείς να δραστηριοποιηθεί με ένα και μόνο e-shop σε ολόκληρη την Ευρώπη τουλάχιστον, όχι με νόμιμο τρόπο. Και αυτό σας το λέω μετά από 20 χρόνια εσωτερικής αγοράς και σχετικής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. Δηλαδή πραγματικά είναι ε, ε, αρκετά μεγάλη αυτή η αποτυχία. Και πράγματι θα πρέπει κάτι να γίνει εδώ, είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι. Άρα λοιπόν μία τέτοια πρόταση οδηγίας ε, αποτελεί ένα μικρό βήμα προς τα μπροστά, αλλά υπάρχει και κριτική, υπάρχουν και επιφυλάξεις και θα τις ε, παρουσιάσω. Να εξετάσω λοιπόν τώρα και να παρουσιάσω ε, τα προβλήματα, τα επιμέρους προβλήματα. Καταρχήν τεχνικές ασάφειες σε ό,τι αφορά τον, την έννοια του καταναλωτή. Υπάρχει μια απόφαση του δικαστηρίου που αναφέρεται ε, σε καταναλωτές με ε, διπλή ιδιότητα. Δηλαδή ως ιδιώτη και ως επιχειρηματία, για παράδειγμα αγορά ενός οχήματος με διπλή χρήση. Ε, και εκεί είχε με την ομολογία του το δικαστήριο Ταχτή υπέρ ε, της ε, αστής νομοθεσίας ε, που υπήρχε διεθνώς σε αυτό το επίπεδο, ότι δηλαδή η οδηγία με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να έχει μια ανητική επίπτωση. Η πρόταση εδώ δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένα και το non-paper, το οποίο είδα εγώ προχθές, αναφέρει ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να παραμένει στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων. Ο νομοθέτης δηλαδή μπορεί να αποφασίσει να μην εκδώσει σχετική απόφαση, ενώ θα αποτελούσε ευκαιρία να κάνει κάτι τέτοιο. γιατί ε, και τα κράτη-μέλη, ως προς και την έννοια του επιχειρηματία, ε, δεν έχουν μια κοινή στάση ως προς τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες μπορεί να είναι πολύ δικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως δεν είναι ε, με στόχο το κέρδος. Για παράδειγμα, εθελοντικές εργασίες, ψυχαγωγία, χόμπι και ούτω καθεξής από εκεί και μετά εγώ δεν θέλω να προσπαθήσω. Αυτό προσπαθούν ε, κάποιοι συχνά. Να ε, ασκήσω κριτική σε κάποιους ε, κανόνες οι οποίοι δείχνουν να είναι λίγο παράλογοι μέσα στο κείμενο της οδηγίας. Κάποιος προσπάθησε να μου πουλήσει ένα μπαλόνι στο δρόμο. Ε, προηγουμένως και είχα την αίσθηση ότι ενδεχομένως θα χρειαζόταν να συμπληρώσω ένα έγγραφο εκεί και να το υπογράψω για να μπορέσω να αγοράσω αυτό το παρόν. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά είχα αυτή την αίσθηση. σε ό,τι αφορά το πού επικεντρώνεται η υποτική συζήτηση, σε ό,τι αφορά το επίπεδο προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Δεν θέλω εδώ να αυλύνω τη συζήτηση, αλλά ο κατάλογος των σημείων ε, στα οποία παρατηρείται μεγάλη απόκληση από την ισχύουσα νομοθεσία, για παράδειγμα στα κράτη-μέλη, δεν είναι τόσο. Ε, δηλαδή πραγματικά είναι κάποια σημεία με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, τα οποία μπορούμε να επιλύσουμε. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις ε, προθεσμίες παραγραφής ή άλλες αντίστοιχες προθεσμίες. Το δικαίωμα επιλογής Επίσης, δηλαδή το ποιος αποφασίζει στην περίπτωση μιας αγοράς ε, ε, εάν ε, υπάρχει και υποχρέωση σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και ούτω καθεξής. Ή για παράδειγμα στη Γερμανία έχουμε πωλήσει μέσω eBay οι οποίες με βάση τον τρόπο που έχει διατυπωθεί αυτή τη στιγμή η πρόταση οδηγίας δεν περιλαμβάνουν. Δεν περιλαμβάνουν αυτές τις πωλήσει μέσω eBay. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν όλα αυτά τα επιμέρους σημεία, πραγματικά εμπιστεύουμε πλήρω στο bargaining αυτό το δουν και να βρει που λαμβάνει η χώρα ε, στο επίπεδο του νομοθέτητος ώστε να βρεθεί μια λύση. Ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει περισσότερο ο νομικό κλάδο είναι αυτά τα side effects, αν θέλετε, τα οποία θα λάβουν χώρα εκτό του ίδιου του τομέα που καλείται να καλύψει η πρόταση οδηγία. Να αναφέρω και πάλι εδώ κάποια παραδείγματα. Προθεσμίε παραγραφή ή άλλε συγκεκριμένε προθεσμίε. Στην Αγγλία, σύμφωνα με ένα στάτιο έχουμε 5 χρόνια στη Σκοτία, 6 χρόνια προθεσμία για καταναλωτικά αγαθά και με μια τέτοια νέα οδηγία στην Αγγλία θα ίσχυαν μόνο δύο χρόνια παρότι η πρόταση ρητά λέει ότι δεν έρχεται να, να παρέμβει στην εθνική νομοθεσία. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση ένας επιχειρηματίας θα βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα από τον καταναλωτή. Βέβαια εδώ ακριβώς η σύγκριση δεν είναι ε, απολύτως σωστή γιατί βέβαια διαφορετικό το, το δίκαιο στο, στο χώρο του καταναλωτή το οποίο είναι υποχρεωτικό και δεσμευτικό και διαφορετικό το B2B, business to business. Αλλά και εδώ θα πρέπει να γίνει ε, κάτι παραπάνω και να αναφέρω αυτή τη μεταφορά της ε, νήσου η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα, μια θάλασσα χάους. Αυτή η μεταφορά είναι ε, πολύ ωραία για το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αν ε, κοιτάξουμε αυτή τη μεταφορά στο εθνικό επίπεδο, βλέπουμε ένα ε, σπίτι το οποίο είναι χτισμένο με ωραίο τρόπο, είναι ένα πλήρες σπίτι και ξαφνικά έρχεται ένας Ευρωπαίος νομοθέτης, αρχίζει και γκρεμίζει έναν τοίχο εδώ, βγάζει κάτι από εκεί και ό,τι καθεξής. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να, κάνουμε, να συντονιστούμε καλύτερα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ε, το, η κοινοτική νομοθεσία να έχει ανηθική επίπτωση. Συμπεράσματα. Τι μπορούμε καταρχήν να κάνουμε με αυτήν την ε, οδηγία. με τη μορφή που έχει τώρα δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε και δεν μπορούμε να, να έχουμε απλά μια γενική ρήτρα. Ε, για παράδειγμα, ένα άρθρο 4 από το οποίο θα λέει δεν ισχύουν αυτά για τον υπόλοιπο κόσμο και το Όχι, θα πρέπει να ε, τη διατρέξουμε άρθρο προς άρθρο, σημείο προς σημείο αυτή την πρόταση οδηγία και αυτό το non-paper περιλαμβάνει μία σειρά από ρεθίσματα για σκέψη παρότι Βέβαια, χρειάζονται πολλέ περαιτέρω διευκρινήσει. Γίνονται κάποιε αναφορέ στο non-paper, ε, ερμηνεύουν κάποια πράγματα, αλλά ε, δεν ε, είμαστε σίγουροι ότι έτσι αναφέρονται στην πρώτη οδηγία και δεν ξέρω αν το δικαστήριο θα αντιληφθεί με τον ίδιο τρόπο και τι σχετικέ διατάξει. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιε τρίτε οι οποίε να εισάγουν κάποια ευελιξία. Για παράδειγμα, μία αρμοδιότητα των κρατών μελών σε περιπτώσει ανάγκε, όπου δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση και Ένα ακόμα σημείο. Η οδηγία δεν θα φτάσει ε, στο σημείο που επιθυμείτε. Δηλαδή η συζήτηση ακόμα και μετά την έγκριση μιας τέτοιας οδηγίας θα είναι καλύτερη αλλά δεν θα έχει επιληθεί. Δηλαδή και πάλι δεν θα μπορεί κανείς να έχει ένα ενιαίο e-shop το οποίο να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Θα με ρωτήσει κανείς ε, πού βρίσκονται οι διαφορές. Ε, Ήδη όμω αυτό διαφάνηκε από τα ερωτήματα. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να δώσουν περισσότερα δικαιώματα με την εθνική του νομοθεσία τα κράτη-μέλη ή όχι. Και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα προφανώ και θα πρέπει ο, ο πολιτής, ο επιχειρηματίας να, να σεβαστεί αυτά τα δικαιώματα. Ε, και εδώ έρχεται τώρα και το ενδιαφέρον σημείο. Θα πρέπει να έρθει ε, με περισσότερε προτάσει, με νέε προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το ε, βασικό λοιπόν ερώτημα εδώ, το θεμελιώδε ερώτημα που με ενδιαφέρει είναι το κατά πόσο επιθυμούν τα θεσμικά όργανα που νομοθετούν να υπάρχει μια τέτοια ρύθμιση ε, με, πρόταση, με οδηγία. Εγώ θεωρώ λοιπόν πως αυτή η μερική, η επιλεκτική εναρμόνιση είναι λανθασμένη. Είτε δηλαδή δεν είχε το θάρρος να περιοριστεί ακόμα περισσότερο, είτε δεν είχε το θάρρος να έχει μια πιο ευρεία εναρμόνιση, να προτείνει μια ευρύτερη εναρμόνιση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί πάντω μια πρόταση όπω έχει τώρα. σω θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι στο πλαίσιο του προγράμματο του Στοχόλμη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να υπάρξει ένα μη δεσμευτικό νομοθέτημα. Νομίζω πω κάτι τέτοιο θα είχε τι ε, ε, λιγότερες δυνατές αμυντικές επιπτώσεις θα ήταν η λύση η οποία θα ήταν η, πιο, η πλέον εγκύτερη στην αγορά και θα ε, σεβόταν με τον καλύτερο τρόπο την ε, λειτουργία της και τα δικαιώματα των συμμετοχών στην αγορά. Αυτά γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να υπάρξουν προβλήματα. Νομίζω πως αυτό το τόνισε επανειλημμένα στην ομιλία μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Well, thank you very much indeed. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή. Έγραψα πολλά πράγματα από αυτό που είπατε, γιατί ακούσαμε διάφορα ενδιαφέροντα, ειδικά όσον αφορά την τεχνολογία. Και είναι αλήθεια ότι ακόμη και εγώ που είμαι μηχανικός ε, δεν τα κατάλαβα τόσο καλά. Δεν ξέρω τι κατάλαβαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εν πάση περιπτώσει έχουμε περίπου ένα τέταρτο στη διάθεσή μας για ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος είναι αρκετά γενναίος για να κάνει ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Βλέπω την κυρία Γκέπχαρντ. Τη βλέπω έτοιμη και θαραλέα να ξεκινήσει την εξέταση, ανάκριση. Absolut nicht, ε, δεν θέλω εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, Πρόεδρε. Απλά θέλω να αντιληφθώ καλύτερα τι ε, τελικά καλούμαστε να καταφέρουμε ως νομοθέτη και τι, ποιο είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό άλλωστε είναι και ο στόχο τη σημερινή ακρόαση. Ε, κύριε ε, Σούντερ Νόλκε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. στο τρίτο σημείο, είπατε πως για σας ε, το τρίτο αυτό σημείο δεν είναι τόσο σημαντικό για σας, αλλά για μας είναι το πλέον σημαντικό, δηλαδή προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αυτό συζητείται πάνω απ' όλα, μαζί με το ζήτημα του κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε πλήρη ή μη πλήρη, μερική δηλαδή εναρμόνιση. Αναφερθήκατε σε τρεις τομείς. Προθεσμία παραγραφής, δικαίωμα επιλογής, σε ό,τι αφορά ε, αντικατάσταση ή επισκευή και πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Πρόκειται για τρία πάρα πολύ σημαντικά σημεία που άπτονται της προστασίας των καταναλωτών. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω και πάλι σχετικά με ένα ε, σημείο το οποίο δεν αντιληφθήκα απολύτω. Τι ακριβώ εννοείται όταν λέτε side effects, παρενέργειε εντό εισαγωγικών. Και είπατε πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν, ε, είτε δεν επέδειξε το απαραίτητο θάρρο, είτε ήταν υπερβολικά θαραλέα. Τι ακριβώ εννοείται με αυτό, γιατί θα ήθελα να λάβω ε, περισσότερε πληροφορίε ε, καθώ δεν με βέβαια ότι έχω αντιληφθεί πλήρω το τι εννοούσατε. Σα ευχαριστώ. The rapporteur Και ο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε, τον Κύριο Σουλτονόλου για αυτή την ε, σαφή και ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Είχα θέσει και προηγουμένω ένα ερώτημα το οποίο απαντήσατε για λόγου σαφήνεια θα ήθελα να το διευκρινίσω. Ποιο είναι λοιπόν το ε, όφελο του να αναφέρει η, ε, στην πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θίγεται η εθνική νομοθεσία. Ε, γιατί νομίζω πως ο στόχος της πρότασης θα ήταν ακριβώς για τους επιχειρηματίες ε, ότι θα υπάρχει πλέον εναρμόνιση, πλήρης εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ε, τότε δεν επιτυχάνουμε τον στόχο που είναι και ταυτόχρονα την μεγαλύτερη ενημέρωση ό,τι αφορά τα δικαιώματα. Ε, και επίσης, ένα ακόμα σημείο θα ήθελα να θίξω, Συζητείτε επανειλημμένα ε, στην, ε, ε, στην, στην κοινή γνώμη η, ο συγκεκριμένο περιορισμό δικαιωμάτων, δηλαδή με μία κίνηση. σω επειδή αναφερθήκατε και εσεί σε αυτό, μπορείτε να μα δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα. Να, μην λέμε δηλαδή, να μην είμαστε γενικόλογοι και να λέμε απλά ότι χειροτερεύει τα πράγματα αυτή η πρόταση. Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ ο Σούλτον Ενόλ και ε, επιβεβαίωσε κάποιε από τι ανησυχίε τι οποίε είχα ήδη κατά την τελευταία συζήτηση τονίσει, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που αναφερθήκατε ότι δηλαδή αυτή η εστιασμένη τελικά αναρμόνιση δεν είναι ε, ο σωστό δρόμο. Αλλά τελικά αυτό εξαρτάται από το ποια είναι τα σημεία εκείνα τα οποία αποφασίσουμε να, να Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι δυνατό ότι κάποια συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία επιλέγουμε να εναρμονίσουμε να, τελικά να μας βοηθήσουν. Ε, και θεωρώ πως ε, τα κράτη-μέλη ε, θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να μην εφαρμόσουν ή τουλάχιστον να μην παρεκκλίνουν από τα όσα ήδη ισχύουν και τελικά να οδηγηθούμε σε μια περίπτωση ότι κάποιο δεν επιθυμεί τίποτα και κανένα δεν επιθυμεί κάτι, αλλά τελικά να έχουμε μια κοινή συμφωνία και μετά τι να πούμε, ότι για παράδειγμα θα υπάρξουν κάποιε ελάχιστε προθεσμίε, τι οποίε θα καλούνται να εφαρμόσουν όλοι αλλά θα υπάρχουν ταυτόχρονα και ανώτατα όρια. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν, αν θέλετε, τα όσα θα ισχύουν, ούτως ώστε να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο ένα κομμάτι τουλάχιστον με μια μερική εναρμόνιση. Κύριε Άριας, σας Παρακαλώ, ε, αν θέλετε να είστε σύντομο, εγώ βλέπετε είμαι αρκετά επίκη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, βεβαίω και θα είμαι πολύ σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή για την ευκαιρία ε, που μου δίνει να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είχα αναφερθεί και προηγουμένω. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πράγματι ότι ο, καταναλωτής στο διαδίκτυο δεν προστατεύεται καθόλου. Γιατί αυτό εξαρτάται από ε, τον, από το, ε, τον, τα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία ποτέ δεν είναι ξεκάθαρα. Να σα πω λοιπόν, δεν συμφωνώ με την απάντηση τη Επιτροπή, γιατί πιστεύω ότι στην οδηγία δεν αναφέρεται καθόλου, ε, η, καθόλου ε, η αγορά μέσω διαδικτύου. Και δεν γίνεται καμία αναφορά σε σχέση με την ε, δυνατότητα αγωγής του, του καταναλωτή και με τις εγγύησεις. Και δεν μου απάντησε σε αυτό που είπα, να δημιουργήσουμε δηλαδή αυτή την ευρωπαϊκή ε, εγγύηση για τις αγορές μέσω διαδικτύου. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για να είμαστε και δίκαιοι, είπε η Επιτροπή ότι αυτό που ισχύει για τις πωλήσει εξ αποστάσεως ισχύει και για τις αγορές διαδικτύου. Αλλά, κοιτάξτε όμως, εσείς είπατε ότι Τώρα το θέμα ποιο είναι. Τα, τα, πώς, πώς, πώς διέπονται νομικά ε, τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Και ε, το ξέρουν οι εταιρείε ότι δρούν ε, πολλές φορές παράνομα ε, και υπάρχει πιθανότητα δίωξης. Τι ακριβώς γίνεται. I think I'll give you the floor then, Professor. Ο λόγος σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ε, ελπίζω να πρόλαβα να σημειώσω τις περισσότερες από αυτές. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα που έθεσε ο Πρόεδρος. Ε, ε, το πρόβλημα της δημιουργίας ενός e-shop το οποίο θα ισχύει για όλη την Ευρώπη και θα είναι νόμιμο είναι ένα πρόβλημα των πολιτών. Γιατί υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία το οποίο εφαρμόζουν με σωστό τρόπο τις δικέ του διατάξεις και μετά βρίσκονται τελικά δηλαδή να δέχονται όλα αυτά τα πειρά όσοι προβαίνουν σε αυτές τις ε, πωλήσει. Ε, βέβαια γνωρίζω ότι θα ακούσουμε περισσότερα από άλλου εμπειρογνώμονε εδώ, οπότε δεν θέλω εδώ να προδικάσω τα όσα γνωρίζουν άλλοι με τη δική του εμπειρία. Αλλά ε, σε ό,τι αφορά το σήμα υπάρχει ήδη, αλλά θα πρέπει να κάνουμε εδώ μια διαφοροποίηση ανάμεσα στου τρει ε, τομεί, για του οποίου μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο σήμα. Καταρχήν για τα προϊόντα, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να αποτελεί αρμοδιότητα του νομοθέτη. Ένα σήμα ποιότητα σε, σε ό,τι αφορά ένα e-shop, δηλαδή το ότι προβαίνει γρήγορα στι ε, προμήθειέ του, ότι φέρεται με το σωστό τρόπο και ούτω καθεξή. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Και αυτό μπορεί να τον έλαβε η αγορά. Αλλά υπάρχει, υπάρχει και δυνατότητα που θα ήταν ενδιαφέρουσα να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομικό σήμα και να υπάρξει για παράδειγμα δυνατότητα ενός πρόσθετου εργαλείου. Ε, κάτι το οποίο θα προωθεί την εσωτερική αγορά και ταυτόχρονα θα αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Δηλαδή ένα σήμα ποιότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι τέτοιο ενδεχομένω να ανταποκρίνεται και στον, ε, στην πρόθεση του Ευρωπαίου νομοθέτη. Δηλαδή να γίνεται κάτι τέτοιο ορατό και να φαίνεται και στα ίδια τα ΙΣΟΒ. Κύριε Λέχινα, η ιδέα αυτών των ε, ελάχιστων, ε, δηλαδή κατώτατων και ανώτατων ορίων, χωρίς να υπάρχει ακριβής εναρμόνιση, ε, να έχουμε απλά ένα περιθώριο αν θέλετε και αυτό δεν είμαι τόσο σίγουρος. Για παράδειγμα να σας, να σας πω το εξής, θέλετε εσείς να δημιουργήσετε ένα e-shop και έχουμε ένα κατάλογο με 100-150 σημεία τα οποία θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη δημιουργία αυτού του e-shop του ηλεκτρονικού καταστήματος διαδικτυακού. Α, ζητώ συγγνώμη, λέω και ξέχασα να κατά κάτι από τον κύριο Άρε. Έχουμε λοιπόν 50, 60, 70 σημεία στα οποία διαφοροποιείται η κατάσταση και όπου θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας αυτές τις διαφοροποιήσεις. Ε, εάν λοιπόν περάσει μια οδηγία η οποία θα έχει αυτά τα ανώτατα 100 τα όρια, ναι, από, αντί για 150 σημεία θα έχετε λιγότερα, θα έχετε περίπου το τρίτο ενδεχομένω, αλλά παρόλα αυτά θα παραμείνουν σημεία, δεν θα εξαλειφθούν. Ε, Και αντιλαμβανόμαστε γιατί εδώ δεν υπάρχει ε, μεγάλη αναφορά σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και νομίζω πως ο συνάδελφος ε, ε, Γιουζέπε ανέφερε κάτι τέτοιο, δηλαδή ποια είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στα όσα προβλέπει η Ρώμη 1. και τα όσα θα προβλέπει πιο συγκεκριμένα η εν λόγω ε, οδηγία. Δηλαδή το πακέτο, αν θέλετε, αυτά που θέλουμε να καλύψουμε, ναι καλύπτονται, αλλά το κατά πόσο ε, ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε. Θα προσπαθήσω τώρα να απαντήσω πολύ γρήγορα στα ερωτήματα του εισηγητή που ε, κατά κάποιο τρόπο επικαλύπτονται με τα όσα ρώτησε η κυρία Γκέπχαρτς. Ε, προστασία του καταναλωτή. Πού βρίσκονται οι διαφορέ και πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο. Εγώ δεν ήθελα να πω πώ είναι ένα τομέα ο οποίο δεν είναι σημαντικό. Ε, προφανώς ε, θέλουμε εδώ τα καλύτερα να επιτύχουμε, δηλαδή τι καλύτερες δυνατές προθεσμίε και ούτω καθεξή. Απλά είπα πως ε, ε, ε, ο αριθμός των σημείων, των επιμέρους σημείων στα οποία υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι τόσο μεγάλος. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την προεδρεσμία, αν αυτή θα είναι δύο χρόνια, όπως βλέπετε στην πρόταση, ή έχουμε άλλη προθεσμία σε άλλα κράτη-μέλη που ενδεχομένως σχετίζεται με το κύκλο ζωής του προϊόντα, δεν είναι κάτι τόσο προβληματικό. Γιατί οι ζημιές, τα ελαττώματα, γίνονται ορατά κατά την πρώτη περίοδο, δηλαδή και όσο με την πάροδο του χρόνου μειώνεται ο, ε, μειώνεται αυτή η πιθανότητα, δηλαδή το κατά πόσο τελικά ένα λάτωμα υπήρχε από την αρχή και διαπιστώνεται στο 5ο ή έκτο ο έτος ε, χρήσης του προϊόντος είναι κάτι το οποίο αμφισβητούμε. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι τόσο δύσκολο θα πρέπει δηλαδή από οικονομική σκοπιά να ε, εξεταστεί κάτι τέτοιο, να δούμε δηλαδή ποια είναι η κατάλληλη προθεσμία. Ενδεχομένω θα πρέπει να γίνεται μια διαφοροποίηση. Υπάρχει διαφοροποίηση, για παράδειγμα, στην ε, πρόταση ε, σε ό,τι αφορά τα κατασκευαστικά υλικά στο δημοτικό δίκαιο. Ίσως εκεί δηλαδή, παράδειγμα, να αποδειχθεί και εκ των υστέρων ε, μετά από ε, μεγάλο διάστημα ότι πρόκειται για ελαττωματικά προϊόντα. Μετά, ε, ήταν ε, το άλλο σημαντικό ερώτημα που θέσατε το τι νόημα έχει να έχουμε αυτό το εναρμονισμένο νησί εάν εκτός αυτού του νησιού, δηλαδή σε όλο εκείνο το, τη θάλασσα παραμένει το χάος και παραμένουν όλες αυτές οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και μπορούν να δημιουργηθούν και νέες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εάν παραμένουμε σε αυτό τον κατάλογο που ανέφερα στη λίστα, όπου ε, τα σημεία εκείνα που βρίσκονται πάνω στο νησί, ναι, εντάξει, επιλύονται, αλλά απλά μειώνεται ο αριθμό των ε, προβλημάτων, δεν εξαλείφεται ο αριθμός. Και άλλωστε μπορούν αυτά να μετατεθούν όλα αυτά τα προβλήματα στο γενικό ενοχικό δίκαιο με αποτέλεσμα τελικά ο αριθμός των προβληματικών σημείων και πάλι να αυξηθεί. Άρα λοιπόν ίσως πραγματικά να ήμουν λίγο κατηγορηματικός όταν είπα ότι είναι λανθασμένη η κατεύθυνση που ακολουθούμε αλλά πραγματικά αμφισβητούμε το κατά πόσο ε, μια τέτοια ε, μερική εναρμόνιση ε, έχει υπερβολικά υψηλό αντίτιμο στο επίπεδο δηλαδή της αποδιοργάνωσης αν θέλετε της εθνικής νομοθεσίας σε αυτούς τους τομείς. Άρα λοιπόν οι εναλλακτικέ είναι είτε μεγαλύτεροι, ευρεία εναρμόνιση ή μερική μη δεσμευτική, μη δεσμευτική εναρμόνιση που έρχεται συμπληρωματικά με δικαίωμα δηλαδή επιλογής για τα με Κυρία Γεύχαρη, νομίζω πως εν μέρη τουλάχιστον απάντησα στο ερώτημα σας. Το ένα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τι συμβαίνει με αυτά, ε, με αυτά τα side effects της ε, πανέργειας και κατά πόσο τελικά ε, τι εννοούσα όταν έλεγα δεν ήταν αρκετά θαραλέα, ήταν υπερβολικά θαραλέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, βασικά, ουσιαστικά με αυτό που κάνουμε με, με την κάλυψη αυτών των πολίσεων είναι η μετατόπιση αυτών των ε, στοιχείων από την μέχρι τώρα οδηγία στην, σε αυτή τη νέα. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή είναι τα μοναδικά στοιχεία αυτά τα οποία θα πρέπει να εναρμονιστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ολόκληρη διαδικασία και αυτή εδώ είναι μια διαδικασία Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή την ευκαιρία, καθώς έχουμε και την νέα βουλευτική θητεία του Κοινοβουλίου, να εστιαστούμε το κατά πόσο αυτή η τετριμένη, αν θέλετε, αυτός ο τετριμένος στόχος μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο ή ε, με, τόσο, ε, με τέτοια ταχύτητα. Ίσως να χρειαζόμαστε άλλα 10-15 χρόνια για να επιτύχουμε πραγματική εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Η κυρία Τουρέν βρισκόταν στην ε, λίστα, αλλά την δεν την είδα. Έχετε τώρα τη δυνατότητα να ρωτήσετε τον καθηγητή άμα θέλετε. Ναι. Αναφερθήκατε σε ένα είδος ε, έκτακτης ανάγκης αν θέλετε, δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες θα μπορεί να ενεργοποιείται το κράτος. Ε, τι ακριβώς εννοούσατε. Ναι, υπάρχουν κάποια παραδείγματα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες των ε, προϊόντων ή στο, στην νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα σημείο στο οποίο δεν αναφέρθηκα είναι το εξή. Ε, ο τομέας, στον οποίο λαμβάνει η χώρα η πλήρης εναρμόνιση, ε, δεν υπάρχει ε, η δυνατότητα πλέον για τα κράτη-μέλη να αντιδρούν με γρήγορο και ευέλικτο τρόπο σε εξελίξεις στην αγορά. Για παράδειγμα, είχαμε μία περίπτωση αυτού του calling στα, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να να υπάρχουν κάποια μικρά τοπικά προβλήματα και τελικά να πρέπει να ενεργοποιείται ολόκληρη αυτή η τεράστια ευρωπαϊκή νομοθεσία για να επιληθούν τόσο περιφερειακά προβλήματα. Άρα λοιπόν ε, σε ορισμένους ιδιαίτερα δύσκολους ε, τομεί ε, με καινοτόμε δηλαδή εμπορικές πρακτικές θα ήταν ε, λίγο ε, ε, επικίνδυνο να απολέσουν τα κρατη τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να αντιδράσουν στην εξέλιξη στην αγορά. Είναι νομίζω όπως βέβαια αρμοδιότητα και υποχρέωση των κρατών μελών να αναφέρουν κάτι τέτοιο, αλλά είμαι σίγουρος πως θα το, πως θα το λάβουν υπόψη τους ως πρόβλημα. Ευχαριστώ. Um, σας ευχαριστώ για τις πολύ περιεκτικές σας απαντήσεις στις ερωτήσεις. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να μιλήσω για το πρόγραμμά μας. Υποθέτω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σχολιάσει. Θα ήθελα να του ζητήσω να κάνουν ερωτήσεις αφού ακούσουμε όλους τους εμπειρογνώμονες στην ε, τελική συνεδρία με ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους τέσσερις εμπειρογνώμονες που έχουμε προσκαλέσει σήμερα και θα ήθελα να τους ζητήσω να μιλήσουν όχι παραπάνω από δέκα λεπτά. Ε, θα έχουμε και το ηλεκτρονικό ρολόι, παρόλο που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες ε, μετρολογίας που συζητούσαμε το πρωί. Θα ακούσουμε τον κύριο Κάρλος Αλμάρας, υποδιευθυντή του Business Europe, ο οποίος ε, μας είχε επισκεφτεί και τον Απρίλιο, τον κύριο Πιέρ Σαλανσόν, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Forward, της εταιρείας Forward, με συγχωρείτε, και μία μεγάλη φίλη της εσωτερικής αγοράς γιατί έχει έρθει πολλές φορές στην Επιτροπή μας και έχει μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες της η κυρία Μονίκου Αγιάν από το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών ΜΠΕΟΚ. Και τέλος ο κύριος Μπομπ Σμίτς Σύμβουλος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της ε, Ένωσης Καταναλωτών Λουξεμβούργου. Θα δώσω καταρχάς τον λόγο στον κύριο Άλμαρας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κύριο Χάρμπορ και τον κύριο Σφάμπ για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης και τη συνέχιση του διαλόγου με τους καταναλωτές για αυτή τη σημαντική πρόταση. Να σας υπενθυμίσω ότι από την έγκριση της πρότασης το 2008 έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ ενδιαφερομένων μερών για το πώς θα λειτουργήσει η οδηγία στην πράξη. Γνωρίζετε ότι παράλληλα με αυτή τη συζήτηση αρκετές οργανώσεις όπως η Business Europe και η BERC έχουν κάνει έναν άτυπο διάλογο για αυτό το θέμα. Από το διάλογο προκύπτει ότι και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν κοινό συμφέρον να έχουμε μια σαφή νομοθεσία κοινή για όλους η οποία θα βρίσκει την κατάλληλη ισορροπία για όλους. Επίσης, από το διάλογο προέκυψε πόσο πολύπλοκη είναι η πρόταση και πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε τις συνέπειες της και για τα κράτη-μέλη, αλλά και για τους τομείς που καλύπτονται. Η στάση μας παραμένει αυτή της πολύ θερμής υποστήριξης, γιατί η οδηγία δημιουργεί ένα πλαίσιο που θα δίνει σαφείς κανόνες όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο και τους καταναλωτές. Θέλουμε μία οδηγία πλήρους εναρμόνισης με ένα σαφές πεδίο εφαρμογής που θα καλύπτει θέματα διασυνοριακού εμπορίου και άλλα θέματα της εσωτερικής αγοράς. Ήδη ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές τα ωφέλη της οδηγίας, αλλά εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στα ωφέλη για τους καταναλωτές, όχι μόνο στα ωφέλη για την αγορά και τις επιχειρήσεις. Νομίζουμε ότι θα αισθάνονται πιο σίγουροι οι καταναλωτές όταν κάνουν διασυνοριακές αγορές γιατί θα γνωρίζουν ότι θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας από όπου και αν αγοράζουν. Επίσης θα είναι πολύ πιο εύκολες οι διαδικασίες και πιο συγκρίσιμες μεταξύ χωρών. Και βεβαίως και η εσωτερική αγορά και η οικονομία θα επωφεληθούν από αυτή την πρόταση μέσω του καλύτερου ανταγωνισμού που θα υπάρξει τόσο για τις τιμές όσο και για την ε, πρόσβαση σε προϊόντα και σε μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Βεβαίως δεν είναι τέλεια αυτή η πρόταση και χρειάζεται να υπάρξουν αρκετές βελτιώσεις. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει επεξηγήσεις, το ίδιο και το Συμβούλιο σε κάποιο βαθμό. Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε πολλές διευκρινήσεις σε θέματα όπως ε, το πεδίο εφαρμογής και οι ορισμοί, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής. Επίσης, ε, οι συνέπειες για την ε, εθνική νομολογία, ειδικά όσον αφορά το συμβατικό δίκαιο. Επίσης, θέλουμε να γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις στην πρόταση αυτή κατά αυτή, έτσι ώστε όταν μιλάμε για δικαιώματα καταναλωτών να μιλάμε και για δικαιώματα και για υποχρεώσεις. Γιατί ο καταναλωτής είναι ισότιμο μέρος και πρέπει να έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επομένως πρέπει να λειτουργεί με την δέουσα επιμέλεια και ο καταναλωτής και να είναι υπεύθυνος για όποιες ζημιές προκαλεί αυτός. Επίσης, θεωρούμε ότι η ισορροπία αυτή τη στιγμή μεταξύ συμφερόντων καταναλωτή και επιχειρήσεων δεν είναι η κατάλληλη αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ούτε τα υψηλότερα ούτε τα χαμηλότερα στάνταρ που ισχύουν στην εθνική νομοθεσία. Πάντως αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι η ισορροπία κλείνει εις βάρος ε, των επιχειρήσεων. Αναφέρω το ότι ο επιχειρηματίας δεν πρέπει να καλύπτει το κόστος ε, για αποστολή κατεπίγουσα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αναλαμβάνει το κόστος μόνο για αποστολή με κανονικό ταχυδρομείο ή οτιδήποτε άλλη κανονική αποστολή. Επίσης, βλέπουμε ότι ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων για οτιδήποτε εντό 7 ημερών, ακόμη και αν πρόκειται για κάποια ίσονο σημασίας αποστολή σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση αποστολής. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και θέματα ανωτέρας βίας, καθώς και κάποια διαβάθμιση ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας. Επίσης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ε, ελευθερία σύναψης σύμβασης και των δύο μερών η οδηγία. Και για θέματα όπως ε, η παράληψη πληροφοριών, οι εγγυήσει και οι αποζημιώσεις θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα θα αναφερθώ και στο έγγραφο το non-paper που λάβαμε χτες, αν και είναι προκαταρκτικές οι απόψεις μου. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό πρώτο βήμα που δίνει κάποιες διευκρινήσεις για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίες θα είναι πρόσδεκτες. Παρ' όλα αυτά να πω ότι παραμένουν κάποια ερωτήματα για εμάς και ελπίζουμε ότι θα λάβουμε απαντήσεις. Σύντομα. Επίσης, η σχέση με αυτό ταξί αυτής της οδηγίας και την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και άλλες σχετικές οδηγίες πρέπει να φανεί πιο σαφώς, να υπάρξουν περισσότερες επεξηγήσεις από ό,τι έχουμε τώρα. Όσον αφορά τώρα τις συνέπειες ε, για την εθνική νομοθεσία και τα εθνικά ένδικα μέσα. θέλουμε να μάθουμε πώς θα προσαρμόσει η Κομισιόν την πρόταση σε αυτά τα εθνικά ένδικα μέσα. Και ιδιαίτερα θέλουμε να δούμε τι προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για τα εθνικά ένδικα μέσα προκειμένου να μην επηρεαστούν από την οδηγία και επίσης μας ενδιαφέρουν και οι συμβάσεις ημικτές που περιέχουν δηλαδή και υπηρεσία και προϊόν. Πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις εκεί. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το πεδίο εφαρμογής. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ε, ποιες υπηρεσίες καλύπτονται και με ποιον τρόπο. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με συμβάσεις διπλής χρήσης. Σύμφωνα με το non-paper, και τα όσα διαβάσαμε, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, ιδιωτική χρήση και το κατά πόσο η διαφορετική χρήση μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα εφαρμόσετε η σύμβαση. Γενικά χρειάζονται αρκετές διευκρινήσεις, πάντως ζητάμε από την Κομισιόν να μας πει να μας διευκρινίσει ποιες τροποποιήσεις θα αφορούν το διατακτικό και ποιες θα έχουν ε, αντίκτυπο μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις. Τώρα, όσον αφορά το συγκριτικό πίνακα, δίνει μια καλή συνοπτική εικόνα των συνεπειών που θα υπάρξουν γενικά και στις εθνικές νομοθεσίες. Βλέπουμε πάντως ότι η προστασία των καταναλωτών ενισχύεται συνολικά. Άρα ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να μας δώσει διευκρινήσεις και να διανύμεις όσο το δυνατόν περισσότερους εταίρους των non-paper με τις διευκρινήσεις γιατί αποτελεί σημείο κλειδί για τη συζήτησή μας. Επίσης ζητάμε από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις συνέπειες που θα υπάρξουν για όλους τους τομείς της οικονομίας γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ένα προϊόν που θα επιστρέφεται θα είναι πολύ δύσκολο να απολυθεί. Τέλος, όσον αφορά την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Αισθανόμαστε ότι εξετάζεται η πρόταση σε πολύ εθνικό επίπεδο, από πολύ εθνική οπτική γωνία και θέλουμε να αλλάξει αυτή η προσέγγιση γιατί κάτι τέτοιο υποσκάπτει το στόχο της πλήρης εναρμόνισης και δημιουργεί εμπόδια για το ελεύθερο εμπόριο. Τέλος, να πω ότι η Business Europe δεν είναι δογματική. Νομίζουμε ότι και η Κομισιόν έχει αναφέρει κάποια πράγματα που αναφέρουμε και εμείς. Θέλουμε να υπάρξει συζήτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να περιορίσουμε τους στόχους μας για πλήρη εναρμόνιση. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή του Κοινοβουλίου να σκεφτεί ευρωπαϊκά και να λάβει υπόψη της ε, το ευρωπαϊκό συμφέρον. Γιατί μία εθνική προσέγγιση εδώ θα οδηγήσει σίγουρα σε αποτυχία και σε προβλήματα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που μείνατε μέσα στα χρονικά περιθώρια. Τώρα, κύριε Σαλανσόν, θα, Σαλανκόν, θα δείξετε κάποιες διαφάνειες. Ελπίζω να έχουν μεγάλα γράμματα οι διαφάνειές σας, γιατί οι οθόνες είναι μικρές. έχετε μοιράσει και αντίγραφα. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα έχετε πάρει και αντίγραφα των διαφανειών. Έτοιμοι, ωραία. Έχετε το λόγο. Έχετε λοιπόν και την ε, εικόνα και τις διαφάνειες. Ευχαριστώ. Όπως ε, και ο κύριος Φάβετς και εγώ για πρώτη φορά είμαι στο βήμα. Ε, και ε, να σας κάνω πρώτα δύο σχόλια ε, για ε, την Forwerk, μια γερμανική βιομηχανική ομάδα που δημιουργήθηκε πριν από 120 χρόνια στη Γερμανία, στο Βούπερταλ, μεσαίου μεγέθους με ε, μικρέ θηγατρικέ σε 11 κράτη-μέλη, που όμω που προβαίνει τη δύναμη των προϊόντων τη σε, πάρα πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Ο όμιλο Φορμπέρκ ε, διανέμει κατευθείαν στου καταναλωτέ. Ε, χρησιμοποιώντας τα εναλλακτικά, τους διαβλούς ε, πωλήσει εκτό καταστημάτων και όλο και περισσότερο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η πρόταση λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλε επιπτώσει στι δραστηριότητε του ομίλου Φορβέρκ. Θα σα παρουσιάσω ε, τα εξή δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, σα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα του τι σημαίνει ε, de minimis ε, εναρμόνιση για μια επιχείρηση όπω η Forwerk. Δεύτερον, σα δώσω παραδείγματα συγκεκριμένα του αντίκτυπου τη οδηγία στην ε, προστασία των καταναλωτών. Ακούσατε πολλά πράγματα, ακούσατε τι οργανώσεις των καταναλωτών που σα είπαν ότι η πρόταση οδηγία στην ουσία εφαρμόζει την, μια ερωτική πολιτική, εναρμόνιση προς τα κάτω, ε, σαν τις μηχανίες που κουρεύει τον καζόν. Δεύτε, ακούσατε άλλε απόψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δηλαδή προσπαθούμε να ε, δράσουμε με ισορροπία τι επαγγελματικέ οργανώσει που υποστηρίζουν ότι αντίθετα πρόκειται για την πολιτική, πολιτική του ουρανοξύστη. Δηλαδή όλο και προ την προστασία των καταναλωτών. Εγώ λοιπόν θα σας δείξω συγκεκριμένα στοιχεία, συγκρίνοντα σε συγκεκριμένε περιπτώσεις την πρόταση τη οδηγία και του υφιστάμενου ε, ε, εθνικού νόμου στα 27 κράτη-μέλη ελάχιστη εναρμόνιση από πρακτική άποψη. Παίρνω το παράδειγμα των χωρών Μπενελούξ και τη Γερμανία και τη Γαλλίας. Γιατί πρόκειται για μια γεωγραφική ζώνη όπου υπάρχουν πολλέ διασυνοριακέ δυνατότητε, τουλάχιστον για μια επιχείρηση όπω η Φόρβερκ. Στο μέτρο που έχουμε πολύ μικρέ αποστάσει, όπω καταλαβαίνετε, ε, ε, δεν έχουμε πρόβλημα γλώσσα και γενικά παρόμοια ανατροπία και κουλτούρα ένθεν και ένθεν των συνόρων. Η Φόρβεκ, λοιπόν έχει ε, εγκατάσταση σε δύο από αυτές τις χώρες, εγκαταστάσει στη Γαλλία και στη Γερμανία. Έκανε λοιπόν μια σύγκριση των κανόνων σε περίπτωση υπαναχώρηση για τις πωλήσει εκτός καταστήματος. Παίρνω τρεις παραμέτρους, το σημείο ε, από το οποίο ξεκινά η υπαναχώρηση, το, ε, τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος και από πού ξεκινάει η μέτρηση. Λοιπόν, ξεκινάει η προθεσμία για την πώληση εκτός καταστήματο, από πότε, από την ημερομηνία που, που γράφεται στη σύμβαση. Μονάδα μέτρηση, η ημερολογιακή ημέρα και 8 ημερολογικές ημέρες. Αυτό στη Γαλλία. Στη Γερμανία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ε, το σημείο κίνηση είναι η στιγμή που παίρνει τι νόμιμε πληροφορίε, τι νομικέ πληροφορίε ο, ο καταναλωτή. Η μονάδα μέτρηση είναι εβδομάδα και διάρκεια είναι δύο εβδομάδε. Και έχουμε και μια ειδική περίπτωση εάν η πληροφορία η νομική όσον αφορά το δικαίωμα επαναχώρηση δίδεται στον καταναλωτή μετά τη σύναψη τη σύμβαση. Η, μονάδα μέτρηση είναι μήνα και διάρκεια ένα μήνα. Στι χώρε Μπενελούξ ήταν η πρώτη περίπτωση. Στη Γαλλία ξεκινάμε από την ε, παραγγελία, μονάδα μέτρηση η χρονολογική ημέρα, ημερολογική ημέρα και 7 ε, ε ημέρε. Λουξεμβούργο. Ξεκινάμε από την παράδοση, μονάδα μέτρησης ε, χρονολογική μέρα και 15 ημέρες ημερολογικές. Στο Βέλγιο ξεκινά. Το σημείο κίνηση είναι η υπογραφή της σύμβασης. Να μην το συγχαίουμε με την δέσμευση. Ε, εργάσιμη ημέρα, μονάδα μέτρησης και διάρκεια 7 εργάσιμες. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω εγώ είναι το εξής. Είναι λογικό να έχουμε τόσο διαφορετικούς ε, κανόνες σε μια ζώνη όπου υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες για διασυνοριακές πωλήσει. Ένα άλλο παράδειγμα. Δικαίωμα επαναχώρηση εκτός ε, καταστήματος για τις επισκέψεις που ζητά να κάνει ο επαγγελματία στο σπίτι του καταναλωτή. Τέσσερις μεγάλες κατηγορίες κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή που, ε, ε, ε που, που λαμβάνουν υπόψη αν αγοράσει το προϊόν. Αυτοί που εξαιρούν την, την επίσκεψη μόνο για το προϊόν για το οποίο ζήτησε την επίσκεψη. Το Ηνωμένο Βασίλειο με κάποια ιδιαίτερη περίπτωση για τις επισκέψεις που ζητούνται μόνο για, τις, ε, για την ειρηπόθηκο πίστη και την καταναλωτική πίστη και τέλος τα κράτη-μέλη που δεν έχουν τέτοιες εξαιρέσεις και που δίνουν στον καταναλωτή δικαίωμα επαναχώρηση σε όλες τις περιπτώσεις. Ανεξάρτητα με το αν ζητήθηκε η επίσκεψη όχι. Άλλο ένα παράδειγμα. Δικαίωμα υπαναχώρησης εκτός καταστήματος για τα ποσά κάτω των 60 ευρώ. Έχετε και εδώ ε, τρεις κατηγορίες κατομελών. Τα κράτη-μέλη που εισήγαγαν κατόφλι, πέραν του οποίου ο καταναλωτής, κάτω από το οποίο ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα επαναχώρησης, αυτοί που έχουν ένα κατόφλι με υποπροποθέσει. στη Γερμανία δηλαδή θα πρέπει η παράδοση και η πληρωμή να γίνονται άμεσα και τα κράτη-μέλη τα οποία εφαρμόζουν το δικαίωμα επαναχώρηση σε όλες τι περιπτώσεις ανεξάρτητα από το ποσό. Τώρα, όσον αφορά τα διάφορα ε, κατόφυλλα, γιατί δεν είναι ταυτόσιμα σε όλε τι ε, χώρε μέλη, θα δώσω ένα παράδειγμα. Μία επιχείρηση όπω η Forberg, που ε, πουλάει για παράδειγμα ένα άρωμα 30 ευρώ, εκτό καταστήματο, σε 27 κράτη-μέλη, θα πρέπει να δώσει δικαίωμα παραχώρηση σε 17, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη στα 10. Ρωτώ, είναι λογικό, είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Τώρα, για να ασχοληθούμε με την ουσία. όσον αφορά τι επιπτώσει σε εθνικό επίπεδο ε, για την προστασία του καταναλωτή. Θα προχωρήσουμε ω εξή. Θα σας δείξω ένα χάρτη της Ευρώπης με διαφορετικά χρώματα. Πράσινο, εκεί όπου αυξάνεται η προστασία με την, με την ε, οδηγία. Πορτοκαλί, ε, οι χώρε με τι οποίε τίποτα δεν αλλάζει. Και με κόκκινο, οι χώρες για τι οποίε θα μειωθεί η προστασία με την πρόταση οδηγίας. Πήρα ένα πρακτικό παράδειγμα έχουμε μία σύμβαση στις 3 Οκτωβρίου του 2009, την ερχόμενη, το ερχόμενο Σάββατο. Που θα συν... Όλες λοιπόν οι πληροφορίες έχουν δοθεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Ε, η παράδοση 6, την επόμενη Τρίτη δηλαδή, με την πρώτη της οδηγίας, το τέλος της προθεσμίας είναι 19 Οκτωβρίου 2009 τα μεσάνυχτα. Να το αποτέλεσμα λοιπόν, αν συγκρίνουμε την πρόταση οδηγία με την υφιστάμενη νομοθεσία. Στην ουσία, τέσσερι χώρε. σε τέσσερι χώρε. θα μειωθεί η, πραγματική χρονική διάρκεια υπο... επαναχώρησης κατά μία, σε τέσσερι θα μείνει η ίδια και στι 19 υπόλοιπε, η πραγματική διάρκεια του χρονικού διαστήματος επαναχώρηση, επαναχώρησης θα αυξηθεί. Θέτω το ερώτημα. Αυτή είναι πολιτική της μηχανής του γκαζόν. Όχι, αυτή είναι η πολιτική του ρινοξύστη. Το ίδιο πράγμα με τις, ε, ε, ζητούμενες, με τις επισκέψεις που, επισκέψεις που ζητήθηκαν. Σε όλες, με πράσινο, ε, βλέπετε εδώ τα ίδια πράγματα. Ε, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μειωθεί η προστασία του καταναλωτή. Σε πέντε χώρες θα, θα μείνει η ίδια εκεί όπου δεν εξαιρούνται αυτές οι επισκέψει και σε όλε και σε όλες τις η προστασία θα αυξηθεί. Πάλι, λοιπόν, το ίδιο. Πολιτική ουρανοξύστη. Για το κατόφλι, το ίδιο πράγμα. Η πρόταση οδηγία προτείνει να καταργηθεί το κατόφλι και να εφαρμοστεί το δικαίωμα επαναχώρηση εκτό ε, ε, καταστήματο σε όλε τι περιπτώσει ανεξάρτητα από το ποσό. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει σημαντική αύξηση της προστασίας ε, του καταναλωτή σε πολλές χώρες και στα τους πόσους υπόλοιπους. Σε καμία χώρα δεν θα δούμε να μειωθεί η προστασία. Τώρα. Για να δούμε το λεπτό ζήτημα των εγγύησεων. Σας έδειξα το κεφάλαιο 3, τώρα σας δείξω το κεφάλαιο 4. Έχω χρόνο? Ωραία. Εδώ πήρα το παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε και από άλλες ομιλητές. Διάρκεια της εγγύησης ε, λόγω ελαττωματικής κατασκευή, Δύο χρόνια σύμφωνα με την πρόταση οδηγία. Και κοίταξα τι θα γίνει σε εθνικό επίπεδο. Πράγματι, εδώ βλέπουμε ότι τα χρώματα τελείω διαφορετικά. Έχουμε status quo στι περισσότερε χώρες και τρία κράτη όπου σαφώ θα έχουμε μείωση του επίπεδου προστασία μείον τέσσερα χρόνια στην Ιρλανδία, στο μεγαλύτερο μέρο του Ηνωμένου Βασιλείου, μείον τρία χρόνια στη Σκωτία, μείον δύο μήνε στην Ιταλία και δύο χώρε όπου η κατάσταση δεν είναι τόσο σαφή, η Φινλανδία και οι κάτω χώρε. Όπου η διάρκεια εγγύηση εξαρτάται από τη διάρκεια ζωή του προϊόντο. Για την περίπτωση που πήρα εδώ, μια μικρή ε, συσκευή, ηλεκτρική συσκευή, ξεκινάμε από την ε, προπόθεση ότι είναι πιθανό να έχουμε δύο χρόνια εγγύηση. Βλέπετε λοιπόν πώ έχουν τα πράγματα. Στα περισσότερα κράτη έχουμε το status quo. Ε, αντιστροφή του βάρου αποδείξεω για του πρώτου έξι μήνε. Ξέρετε, στου πρώτου έξι μήνε τη περίοδου εγγύηση, ο επαγγελματία είναι αυτό που πρέπει να αποδείξει ότι το αγαθό δεν είχε ελάττωμα στην κατασκευή του. Ότι όταν παραδόθηκε δηλαδή δεν είχε παρουσίαζε ελάττωμα. Το ίδιο θα γίνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Στάτου έξω από την Πορτογαλία. Γιατί οι Πορτογάλοι έχουν επιλέξει να, ε, η αντιστροφή του βάρους αποδείξεως να ε, ισχύει σε όλη τη διάρκεια ισχύως εγγύης, δηλαδή για τα δύο χρόνια. Τελευταίο παράδειγμα και τελειώνω. Το λεπτό ζήτημα του τρόπου αποζημίωσης. Έθεσε το εξή ερώτημα. Εάν ο καταναλωτής μπορούσε αμέσω να ζητήσει την λύση τη σύμβαση σε περίπτωση ελαττωματικού ε, προϊόντο. Με την πρόταση τη οδηγία δεν μπορεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητήσει επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο, τι βλέπετε. Υπάρχουν ορισμένε χώρε που δεν έχουν ιεράρχηση τη αποζημίωση, Πορτογαλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Λετωνία. Εδώ ο καταναλωτή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε τρόπο και τη λύση τη σύμβαση υπάρχει το περίφημο right to reject, ε, δικαίωμα ε, ε, ε, ε απόρριψη στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση το βάρο αποδείξεω βρίσκεται στον καταναλωτή. Για να λύσει τη σύμβαση ο καταναλωτή πρέπει να αποδείξει ότι υπήρξε ε, ε λάθο στην κατασκευή. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Αν το, το λάθο είναι μικρό, το ελάττωμα είναι μικρό, βλέπετε ότι εδώ έχουμε τρει χώρε όπου ο καταναλωτή μπορεί να ζητήσει άμεσα τη λύση τη σύμβαση. Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, σα λέω το εξή. Πρώτα απ' όλα, ε, ο όμιλό μα πιστεύει ότι η πλήρη εναρμόνιση είναι ο καλύτερο τρόπο για να, σημειώ, να σημειώσουμε πρόοδο. Δεύτερον, τουλάχιστον όσο αφορά τι πωλήσει εκτό καταστημάτων, εξ ε, η πρόταση οδηγία επιτυγχάνει πλήρη εναρμόνιση σε πολύ ψηλό επίπεδο προστασία, για να μην μπούμε στο ύψιστο επίπεδο σε σχέση με το εθνικό. Και όσον αφορά την εγγύηση, συνολικά η πρόταση οδηγία διατηρεί το status quo στα περισσότερα κράτη-μέλη. Αυτά ήθελα να πω και σα ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Σαλανκόν. Πολύ καλή η παρουσίασή σας και πρέπει να σας πω ότι Είμαι σίγουρη ότι ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή ε, θα χρησιμοποιήσει τι ε, γραφικέ σα παραστάσει. σω λοιπόν η επόμενη έκδοση τη Επιτροπή ε, θα χρησιμοποιήσει τα ωραία αυτά στοιχεία και τι γραφικέ παραστάσει που μα δώσατε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανεί τι γίνεται. Πολύ ωραία. Χαίρομαι τώρα γιατί θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκουαγέν, η οποία θα παρουσιάσει τη δική τη προοπτική από μεριά του Μπέοκ. Ευχαριστώ. Η Μπέοκ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών. Εκπροσωπούμε 43 από τις πιο σημαντικές οργανώσεις καταναλωτών σε 23 ευρωπαϊκές χώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ γιατί είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Θα ήθελα να πω κύριε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ε, λάβει το λόγο οι ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών, οπότε ίσως θα έπρεπε να με ακούσετε γιατί μπορεί να ακούσετε και κάποια πράγματα που θα σας εκπλήξουν. Δεν έχουμε πολλά λεπτά στην διάθεσή μας, πάντως να πούμε ότι έχουμε και γραπτό στις απόψεις σας. Αν δεν τις έχετε λάβει τις απόψεις σας, μπορούμε να τις στείλουμε με email στα μέλη της Επιτροπής σας. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχάς ε, κάποια θετικά σχόλια και μετά κάποια αρνητικά. Τα θετικά. Επικροτούμε την ιδιαίτερα επικοδομητική προσέγγιση πολλών από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα θεσμικά όργανα. Ειδικά το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολύ καλή δουλειά για την ανάλυση της βάσης της πρότασης. Επίσης, η Τσεχική Προεδρία έκανε πολλά για να διευκρινίσει το περιεχόμενο της οδηγίας. Και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και με οργανώσεις όπως η Business Europe και που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να κάνουμε σχόλια τα οποία ελπίζουμε ότι θα δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης επικροτούμε ιδιαίτερα την ε, προσπάθεια της Επιτροπής, ειδικά του γραφείου της κυρίας Κούνεβα και την ε, ΓΑΜΑ ΣΑΝΚΟ για τις προσπάθειες που έκαναν για την οδηγία. Όμως, παρά τη σκληρή δουλειά, παρά την επικοδομητική στάση, οι τελευταίες εξελίξεις από πλευράς καταναλωτών κάθε άλλο παρά καθησυχαστικές είναι. Γι' αυτό έχω σήμερα το δύσκολο έργο να σας πω ποιες είναι οι ανησυχίες μας σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν περάσω στα δύο βασικά σημεία με τα οποία διαφωνούμε, θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Αυτό το νομοθέτημα είναι πολύ σημαντικό για την νομοθεσία των καταναλωτών και το αποτέλεσμα είναι πολύ περιορισμένο για το φιλόδοξο σχέδιο από το οποίο ξεκίνησε. Αυτό δεν αφορά μόνο τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Αφορά όλες τις πράξεις των καταναλωτών. Από το να αγοράσετε ένα μολύβι με το να αγοράσετε ένα αεροπλάνο. Άρα χρειάζεται ισορροπία μεταξύ προστασίας καταναλωτών και ελεύθερου εμπορίου στην Ευρώπη. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι όλα τα, όλες οι εγχώριες αγορές το να αγοράσετε εφημερίδα ή ένα βιβλίο επίσης θα επηρεάζεται από αυτή την πρόταση, όχι μόνο οι διασυνοριακές αγορές. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι μπορεί να καθυστερήσει η έγκριση, αλλά από τη στιγμή που θα εγκριθεί θα ισχύει για χρόνια ενδεχομένως για δεκαετίες. Άρα είναι πολύ σημαντικό να τα κάνουμε όλα σωστά. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν γρήγορη νομοθεσία, θέλουν νομοθεσία που θα κρατήσει, θα κρατήσει για χρόνια. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την πρόκληση θα πρέπει ο Ευρωπαίος νομοθέτης να είναι πολύ προσεκτικός και να αφιερώσει πολλή ενέργεια. Να γνωρίζει ακριβώς ποιες θα είναι οι συνέπειες της οδηγίας και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Και αυτό καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό επειδή η Κομισιόν προτείνει πλήρη εναρμόνιση. Κάτι που διεισδύει ακόμη περισσότερο στην εθνική νομοθεσία, γιατί θα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό όριο για την προστασία των καταναλωτών, πέρα από το οποίο δεν θα μπορούν να πάνε οι εθνικές νομοθεσίες. Οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί, γιατί θέτεται ένα όριο για τους καταναλωτές και την προστασία τους. Τώρα, περνάω στις επικρίσεις μου. Το πρώτο βασικό είναι η έλλειψη σαφήνειας. Να πω ότι και χθε 24 ώρες πριν από την ακρόαση λάβαμε αυτό το non-paper. Η γραμματεία μας ε, είχε βοηθήσει λίγο, όμως εγώ ως ε, δικηγόρος από με σπουδές νομικής, ως άτομο με σπουδές νομικής έχω μάθει να μην κάνω σχόλια για τις προηγούμενες εκδόσεις. Είχαμε λοιπόν την προηγούμενη εκδόση του Ιουλίου, αλλά τη τελική έκδοση τη λάβαμε τώρα και μάλιστα είναι non-paper. Γιατί non-paper? Λαμβάνουμε πολλές περιφερειακές πληροφορίες, αλλά ποια είναι η αξία τους επ' αυτόν θα αποφασίσουμε για την νομοθεσία. Χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια, χρειαζόμαστε καλή νομοθεσία. Δεν μπορούμε λοιπόν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις να τα βλέπουμε στις αιτιολογικές σκέψεις ή στα non-paper. Πρέπει να αναφέρονται στο σώμα των οδηγιών, στο ίδιο το νομοθέτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πληροφορία, πληροφόρηση και πληροφορίες από εδώ και από εκεί και δεν γνωρίζουμε τι είναι η επίσημη εκδοχή. Όσον αφορά τώρα τον πίνακα, το είπε και η κυρία Τεστόρη ότι πρόκειται για κάτι που βρίσκεται εν εξελίξη. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι εξαντλητικός ο πίνακας. Δεν συγκρίνει όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας με όλη την υπάρχουσα νομοθεσία σε κράτη-μέλη και δεν συγκρίνει δύο βασικά κεφάλαια νομοθεσίας από πλευράς καταναλωτών. Τις προϋποθέσεις πληροφόρησης και τις συμβάσεις Επίσης, κάτι ακόμη πολύ σημαντικό για εμάς. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες για τον πίνακα. Όμως, παρά τις προσδοκίες μας, αυτός ο πίνακας δεν έχει επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη. Είναι μια εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που χρειάστηκε σκληρή δουλειά μεν, αλλά είναι εκτίμηση της Επιτροπής για την θετική αρνητική επίπτωση στην εθνική νομοθεσία. Και αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Δεν είναι επικυρωμένο, δεν είναι έγκυρο κείμενο. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι μόνο οι εθνικές αρμόδιες αρχές μπορούν να γνωρίζουν τον πλήρη αντίκτυπο αυτής της νομοθεσίας στο εθνικό σύστημα. Και το σημείωμα που βρίσκεται δίπλα στον πίνακα μας δίνει κάποιες διευκρινήσεις, αλλά προκύπτουν και επιπλέον δυσκολίες και συγχύσεις και από το σημείο. Οπότε, συνοψίζοντας, ο πίνακας στην σημερινή του μορφή προκαλεί σύγχυση, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμος πρέπει να τον δουλέψετε πολύ περισσότερο προκειμένου να έχουμε μία σαφέστερη εικόνα για το τι αντίκτυπο θα έχει η, Κομισιόν, ε, για το τι αντίκτυπο θα έχει η πρόταση της Κομισιόν. Και περνάω στο επόμενο βασικό σημείο, την εναρμόνιση. Και θα ήθελα να το τονίσω γιατί πολλές φορές έχουν πει ότι έχουμε την αντίθετη άποψη. Η Μπέκ δεν έχει αυτόματη προσέγγιση όσον αφορά την αρμόνιση. Η πλήρης αναρμόνιση μπορεί να αφαιρέσει τα εμπόδια στην, στο εμπόριο και βεβαίως αυτό που ζητάμε δεν είναι το καλύτερο επίπεδο προστασίας καταναλωτών γιατί δεν μπορούμε να ορίσουμε ποιο είναι αυτό. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν γι' αυτό Φιλανδία και Ενωμένο Βασίλειο για παράδειγμα. Όμως θέλουμε ένα υψηλό επίπεδο Ας μην είναι το υψηλότερο επίπεδο. Τι βλέπουμε με αυτή την πρόταση. Έχουμε μεν πλήρη εναρμόνιση, αλλά το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών δεν είναι αποδεκτό. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι με εκπλήσει που ζητάνε οι επιχειρήσεις ακόμη πιο πλήρη εναρμόνιση. Όμως έχουμε πλήρη εναρμόνιση πριν με φάση εκ πρώτης όψεως. Αυτό παραπλανά τις επιχειρήσεις, γιατί νομίζουν ότι όντως υπάρχει πλήρης εναρμόνιση, αλλά όταν καταλήξουμε σε προσφυγή τελικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα αστικά δικαστήρια και την εθνική νομοθεσία που μπορεί να πάρει χρόνια. Άρα αυτή η διαδικασία είναι παραπληκτική για τους επιχειρηματίες και δεν είναι ο σωστός τρόπος να τους δείξουμε ότι αφαιρούμε τα εμπόδια. Άρα από τη μία πλευρά δεν έχουμε αρκετή προστασία των καταναλωτών, παρόλο που υπάρχουν και κάποιες βελτιώσεις, αλλά για ορισμένες διατάξεις βλέπουμε μείωση της προστασίας των καταναλωτών. Και από την άλλη πλευρά, για τους επιχειρηματίες, δεν έχουμε το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού που θα ήθελαν. Άρα, για εμάς αυτό είναι μία κατάσταση lose-lose. Χάνουν και οι δύο. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχάς, πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο προκειμένου να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα με τις διασυνοριακές συμβάσεις. Πηγαίνετε στο δρόμο οπουδήποτε και ρωτήστε τους καταναλωτές γιατί δεν αγοράζετε διασυνοριακά. Δεν πρόκειται να σας πούνε ότι εξαιτία της νομοθεσίας θα σας πούνε ότι έχουν πρόβλημα με τη γλώσσα και πρόβλημα με την απαστολή προϊόντων. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και όχι ο κατακαιρματισμός της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Πρέπει λοιπόν να βρούμε περισσότερα στοιχεία και να έχουμε ένα καλύτερο, μια καλύτερη ανάλυση αντικτύπου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις και έναν πληρέστερο πίνακα που θα ασχολείται και με θέματα όπως η αστική νομοθεσία κτλ. Δεύτερον, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι πρόκειται αυτή η οδηγία να καλύψει όλα τα θέματα. Όμως, αυτή η οδηγία μπορεί να ισχύει για δεκαετίες, άρα πρέπει να είναι θωρακισμένη για το μέλλον, πρέπει να προστατεύει τον καταναλώτη για την ψηφιακή εποχή. Για παράδειγμα, πρέπει να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τα προβλήματα διαλειτουργικότητας που μπορεί να υπάρχουν για μια ψηφιακή συσκευή. Επίσης, πρέπει να αναφέρονται στους όρους θέματα που έχουν να κάνουν με τις άδειες χρήσης λογισμικού. Αυτά είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα. Τώρα, όσον αφορά το επίπεδο ή τύπο εναρμόνισης ζητάμε εμείς. Και τελειώνω εδώ. Τελευταία πρόταση πάνω Συμφωνούμε εδώ με την προσέγγιση του Κοινοβουλίου που είναι μεικτή. Μπορούμε να έχουμε πλήρη εναρμόνιση σε τομείς όπου υπάρχουν τεχνικά θέματα, όπως για παράδειγμα η περίοδος του δικαιώματος υπαναχώρησης κτλ αν βεβαίως ε, μας εγγυώνται ένα αποδεκτό επίπεδο προστασίας καταναλωτών, αλλά σε άλλα θέματα όπου υπάρχουν είτε εθνικές ιδιαιτερότητες ή όπου εξελίξεις είναι ραχδαίες και πρέπει να μπορούν οι εθνικές ε, αρχές να αντιδρούν άμεσα, εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μία όχι τόσο πλήρη εναρμόνιση προκειμένου να επιτρέψουμε και στις επιχειρήσεις να δουν κάποια εμπόδια να άρονται αλλά και στους καταναλωτές να βλέπουν τα δικαιώματά τους να προστατεύονται. Και να πω ότι εμείς στην ΠΟΙΚ αναρωτιόμαστε μήπως θα ήταν καλύτερο τελικά να ξεκινήσουμε από την αρχή από το να προτιμάμε να κλείσουμε τις τρύπε τώρα. Σας ευχαριστώ για τη σαφέστατη παρουσίασή σας και είχα την εντύπωση, είχα την πρόθεση να πω και σας ευχαριστώ επί τη ευκαιρία για αυτά που είπατε για ε, την προκατοχό μου, την Άλλη Μακάρθη ε, και γνωρίζω και την προηγούμενη ακρόαση ότι και εσείς και η Business Europe συνεργαστήκατε για ορισμένα θέματα και πρέπει να το γράψουμε στα πρακτικά γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τέλος λοιπόν σε αυτό το γύρο για 10 λεπτά ο κύριος Μπομπ Σμίτς από το Λουξεμβούργο. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε κυρίες και κύριοι, η οργάνωσή μου, η Ένωση ε, του Λουξεμβούργου των Καταναλωτών, ανήκει στον ΠΕΟΚ. Γιατί λοιπόν εμείς που είμαστε μικρή χώρα θέλουμε να πάρουμε το λόγο ξεχωριστά. Κυρίως γιατί εξακολουθούμε να είμαστε πρωταθλητές στις διασυνοριακές αγορές. Με περίπου 11% των ετησίων δαπανών, ε, καταναλωτικών δαπανών να προέρχονται από αυτό τον τομέα. Είμαστε λοιπόν μια χώρα που οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες ε, γνωρίζουν ιδιαίτερα τι σημαίνει αυτή η εσωτερική αγορά. Με ε, τα προβλήματα ε, που προέρχονται από τον κατακαιρματισμό της νομοθεσίας. Λοιπόν, μια χώρα τα γνωρίζει όλα αυτά, είναι η δική μας χώρα. Και γιατί αγοράζουμε πέραν των συνόρων. Ε, συγγνώμη, δεν θέλω να ε, περιευτολογήσω γιατί γνωρίζουμε περισσότερε γλώσσε από του υπόλοιπου. Και από την άλλη, είμαστε κάπου στη μέση όσον αφορά την κουλτούρα. Ε, έχουμε μια νοτροπία, ευέλικτη, ευέλικτη αν θέλετε. Είμαστε κάπου ανάμεσα στου Γερμανού και στου Γάλλου. Τέλο πάντων, όλα αυτά μα οδηγούν σε αυτή την παρέμβαση. Κοιτάξτε, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομο γιατί σα έστειλα δύο έγγραφα. Ένα στα αγγλικά, το οποίο είναι βασικό σημείωμα και από το, από το έγγραφο αυτό θα αναφερθώ σε ένα, δύο, τρία σημεία και ελπίζω η Επιτροπή σας να έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει το περιεχόμενό του γιατί εκεί αν θέλετε περιγράφουμε στι λεπτομέρειε τις σκέψεις μας για την πρόοδο που έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σε αυτή την πρόταση οδηγία και ε, ε, έχω και ένα speaking note στα γαλλικά όπου εκεί θα αναφερθώ ε, με δύο λόγια σε αυτά τα οποία αναφέρθηκε η πρόσωπος της Επιτροπής σε σχέση με το δικό σας ανεπίσημο έγγραφο, στο έγγραφο εργασίας. Πολύ σύντομα λοιπόν, όσον αφορά ορισμένα ε, βασικά σημεία του σημειώματο στα αγγλικά. Κανεί δεν το είπε ακόμα, αλλά η πρόταση τη Επιτροπή ε, έχει ξεκινήσει ε, σχεδόν εδώ και ένα χρόνο. Και παρόλο που το Κοινοβούλιο για του δικού του λόγου έχει ξεκινήσει σιγά σιγά, σε επίπεδο Ευρώπη, Επιτροπή Περιφερειών, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, υπάρχει γνωμοδότηση ομόφωνη πλην ψήφου. Ομοφωνία λοιπόν ανάμεσα στα κόμματα και στι και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν μιλάμε για πλήρη εναρμόνιση, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει όλο και λιγότερο περιθώριο αξιολόγηση των εθνικών νομοθετών. Και αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε για εμά του υπόλοιπου, του καταναλωτέ. Γιατί βλέπουμε ότι όσον αφορά αυτά τα δύο κοινοτικά όργανα, αλλά και τα εθνικά, ε, αναφέρομαι στο, ε, στα νομοθετικά σώματα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλία, του Ελληνικού, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, της Γερμανίας, όλοι κατέληξαν σχεδόν ε, ομόφωνα στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή ότι πρέπει, αν πραγματικά θέλουμε να ε, καταλήξουμε στο ζήτημα αυτό, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά η μεικτή προσέγγιση, mixed approach. Δηλαδή, το αντίθετο από αυτό που είπε ο καθηγητής, ορισμένοι τομείς και το Συμβούλιο εξάλλου κατέληξε σε αυτό το στάδιο στο ίδιο συμπέρασμα. οι ορισμοί, η υποχρέωση πληροφόρησης, ένα ζήτημα και από την άλλη, αντίθετα με αυτά που ακούσαμε, όσον αφορά το, τη διάρκεια του δικαιώματος υπαναχώρησης, μπορούμε να φτάσουμε αρκετά μακριά. Δεν ξέρω αν θα πρόκειται για το τέλος του τρόμου. Πάντως ε, κατέληξαν όλοι όσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής ότι σε αυτούς τους τρεις τομείς με λίγη καλή θέληση μπορούμε να καταλήξουμε. Άρα πεδίο εργασίας, τι απομένει. Και εδώ το Συμβούλιο θα δούμε τι θα κάνει. Και ε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για τι εργασίε τη Τσεχική Προεδρία και τη Σουηδική Προεδρία. Τώρα έχουμε το θέμα τη ε, αποζημίωση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντο και στι καταχρηστικέ ρήτρε. Εδώ πρέπει να δούμε πού μπορούμε, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Προσωπικά και τώρα αναφέρομαι στο σημείο τη Επιτροπή. Νομίζω ότι το σημείο τη Επιτροπή στην ουσία παραδέχεται αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε και το οποίο αναφέρθηκε, δεν το επαναλάβω, ότι θα είναι δηλαδή ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξει διασαφήνιση και νομική βεβαιότητα σε επαρκή βαθμό ανάμεσα δηλαδή στο τι θα αποτελέσει αντικείμενο πλήρους εναρμόνισης και στο τι θα ε, παραμείνει σε άλλες νομικές βάσεις, αστικό δίκαιο κτλ. Και ε, σα το λέω ότι όλα αυτά δεν θα διευκολύνουν το έργο ε, ε τη ερμηνεία που θα δώσει το δικαστήριο. Γιατί θα αισθανθεί ε, μεγάλη δυσκολία το δικαστήριο. Ενώ σήμερα με βάση τα άρθρα τη συνθήκη, ελεύθερη κυκλοφορία ε, προϊόντων κτλ. Ε, υπάρχει γνώση για το κατά πόσο το α ή το β μέτρο προχωρεί περισσότερο από ό,τι θα δικαιολογούσε η οδηγία de minimis. Εδώ λοιπόν πραγματικά δυσκολεύουν τα πράγματα ε, και δυσκολεύει ιδιαίτερα ο ρόλος του δικαστή. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι πρέπει να σταματήσουμε όλες τις εργασίες? Όχι, δεν θα ε, έφτανα στο σημείο στο οποίο έφτασε η Μονίκ. Νομίζω ότι προσωπικά, όπως και ο καθηγητής, πιστεύω ότι μπορούμε να σώσουμε ε, τα πράγματα και την κατάσταση. Ας προσπαθήσουμε όμως πρώτα να βελτιώσουμε την ελάχιστη εναρμόνιση. Αξίζει τον κόπο. Ε, κυρίως όσον αφορά τις ε, νομικές εγγύσεις και τα χρηστικές ρήτρες, πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα ακόμα και σε επίπεδο, σε ελάχιστο επίπεδο. Η, η Μονίκ το είπε, πρέπει να φτάσουμε σε μια κατάσταση win-win που να κερδίζουν όλοι. Γιατί, να πάρω το παράδειγμα ε, των εγγύσεων και των ένδικων μέσων. Και εδώ η κυρία Τεστόρη επιβεβαίωσε αυτό το οποίο είπε και η κυρία Κούνεβα πριν από λίγους μήνες στην προηγούμενη ακροασή σας αν καταφέρουμε σε όσο είναι το ψηλότερο επίπεδο, για παράδειγμα, ε, προσθέτοντα και το right to reject, το δικαίωμα ε, λύση τη σύμβαση, να δούμε πού θα φτάσουμε. Και αν τελικά τα κράτη-μέλη φτάσουν σε ένα επίπεδο που δεν είναι επαρκέ ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πλήρη εναρμόνιση, πάντως Ακόμα και εκεί που θα φτάσουμε, αυτό είναι κεκτημένο για όλου και για τι επιχειρήσει. Γιατί σε, περίπτωση διαφωνία, το επίπεδο προστασία του καταναλωτή θα έχει αυξηθεί σε λογικό επίπεδο, άρα λιγότεροι εθνικοί αποκλίνοντα κανόνε κτλ. Η εμπειρία μα πάντω μα δείχνει με σαφήνεια, όπω το είπα, και τελειώνω σε αυτό το στάδιο. Τα υπόλοιπα θα τα θα διαβάσετε, ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε όσον αφορά τα προβλήματα κατακαιρματισμού. Γενικά, η εφαρμογή των εθνικών κανόνων, των διαφορετικών εθνικών κανόνων που υφίστανται στα χαρτιά και πράγματι είναι πολύ διαφορετική αυτοί οι κανόνε αν του εξετάσουμε στι λεπτομέρειέ του. Αλλά πότε τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, όταν οι επαγγελματίε και οι καταναλωτέ δεν μπορούν να βρουν μια λύση μεταξύ του ένα φιλικό διακανονισμό. Όταν λείπει να περάσουμε μέσα από τα δικαστήρια. Ε, τότε οι νομικοί, και εγώ νομικό είμαι, αρχίζουμε να παίζουμε και να βλέπουμε, ε, στο υπόψη το ρωμαϊκό δίκαιο και τα ε, ε, ποια νομοθεσία ισχύει. Ε, τότε φαίνονται τα αποτελέσματα του κατακαιρματισμού. Σε αντίθετη περίπτωση μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά το λεγόμενο κόστος των επιχειρήσεων, δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Στο Λουξεμβούργο, κάθε μέρα έχουμε επιχειρήσεις, πάροχους υπηρεσιών που έρχονται στο Λουξεμβούργο και που καταρχήν σέβονται απόλυτα το δίκαιο του Λουξεμβούργου και χρησιμοποιούν χωρίς το γνωρίζουν καλόπιστα τις γενικές ε, διατάξεις, γενικές προϋποθέσεις, γενικούς όρους, ε, γερμανικούς, γαλλικούς κτλ. Μπορεί να διαφέρουν στο α στο β ε, σε σχέση με αυτά τα οποία ισχύουν στο Λουξεμβούργο. Αλλά σε γενικές γραμμές όλα αυτά δεν δημιουργούν πρόβλημα. Έτσι να τα λέμε τα πράγματα απλά. Και αν υπάρχει ένας κίνδυνος από αυτό το κατακρεματισμό, Τελικά αυτόν τον κίνδυνο θα τον αισθανθεί ε, περισσότερο από όλου ο επαγγελματία. Γιατί εάν δεν καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια βέλγικη επιχείρηση που δουλεύει στο Λουξεμβούργο και είναι διαφορετικό το δικαίωμα επαναχώρηση και πάμε στα δικαστήρια, ε, όλα αυτά γίνονται ορατά ε, και γίνονται, είναι σβάρος της επιχείρησης. Άρα λοιπόν θα σας πω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπο για να σημειώσουμε πρόοδο, στα έγγραφα που ετοίμασα ε, περιγράφουμε την κατάσταση και πρέπει να δούμε και τις εργασίες του Συμβουλίου, κυρίως το ζήτημα αυτό, όχι ε, για κάποιο άλλο λόγο. Όπως είπατε και εσείς ε, κύριε Σουά, πρέπει να έχετε το χρόνο, αλλά κοιτάξτε, ε, αυτή τη στιγμή πρέπει να ενισχύσουμε τα πράγματα. Ο ασθενής δεν πρόκειται να πεθάνει, πρέπει να τον βοηθήσουμε να ζήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και η πρακτική σα εμπειρία σε ό,τι αφορά τις ε, διασυνοριακές συναλλαγές είναι πάρα πολύ πολύτιμη, όπως είδαμε να συμβαίνει και σε σχέση με τις οδηγίε για τις υπηρεσίε και θα σα καλέσουμε και πάλι εδώ ε, σε αντίστοιχε συζητήσει και σα ευχαριστούμε που κάνετε τον κόπο να έρθετε εδώ για να μας ε, κοινοποιήσετε τι απόψει σα και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ε, αναφερθήκατε σε μια νέα μεταφορά. εμεί, μιλάγαμε για νησιά νομικής ε, βεβαιότητας. Τώρα ήρθε η συζήτηση για το μωρό το οποίο θα πρέπει να το σώσουμε το μωρό και να μην το πετάξουμε μαζί με τα, με τα πόνερα όπως ε, έχουμε στα αγγλικά αυτή την ε, παρμία. Τώρα θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στους συναδέλφους μου να θέσουν κάποια ερωτήματα στους εμπειρογνώμονες και στη συνέχεια θα δώσω τη δυνατότητα στον κύριο Ντόλινγκ από την πλευρά δηλαδή του Συμβουλίου να δηλαδή, το λόγο και μετά μπορούμε να κάνουμε γενικότερη συζήτηση. Και βέβαια νομίζω πως θα ήταν δίκαιο και θα συμφωνήσετε να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ε, ε νομίζω πάντως πως θα ήταν καλό να ακούσουμε κάποιες ε, σύντομες συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, στους εμπειρογνώμονες μας. Νομίζω πως ο συγκητής μας θέλει να ρωτήσει μια-δυο να θέσει ένα-δύο ερωτήματα. Κυρία Γκέπχαρτ, Σφάμπ λοιπόν, Γκέπχαρτ, άλλος, ο κύριο Ροσφόρ. Κύριο Σφάμπ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν πολύ χρήσιμε όλε οι παρεμβάσει των εμπειρογνωμών για την περαιτέρω συζήτηση που θα κάνουμε και του ευχαριστώ για αυτό. Και θεωρώ πω οι διαφορετικέ ε, προοπτικές απέναντι σε αυτή την προοπτική έγιναν και αυτές ορατές και νομίζω πως ε, όλοι συμφωνούν, συμφωνούν όπως είπε και ο κύριος Σμίτς πως έχει νόημα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από αυτής της πρότασης. Ταυτόχρονα όμως πως αυτό που είπατε κυρία Γκόγιανς θα πρέπει να ε, είναι τελικά ότι ε, όλα τα στοιχεία αυτής της ε, πρότασης να συμφωνούν μεταξύ τους και να έχουμε μια γενική λύση και να μην έχουμε δηλαδή ένα συνοθήλευμα το οποίο τελικά δεν θα επιλύει κάτι ουσιαστικά. Ε, και να πούμε πως ε, εμείς ε, ως Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θέλουμε να εκπονήσουμε μια μελέτη την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε από κοινού μαζί σας ώστε να μπορέσουμε να την ερμηνεύσουμε και από κοινού. Αλλά κύριε να σας ρωτώ, πιστεύετε πως οι ενώσεις προστασίας των καταναλωτών είναι διατεθειμένες να αποδεχτούν αυτό το στόχο και να ε, συνεργαστούν επικοδομητικά προ αυτόν, δηλαδή για ένα ενιαίο επίπεδο προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή γενικότερα η άποψή του ήταν πω ε, τελικά μια τέτοια, ε, οι επιπτώσει που θα είχε μια τέτοια πρόταση ουσιαστικά είναι αρνητικέ για το επίπεδο τη προστασία του καταναλωτή. Καθώ δεν είναι εφικτή στην υλοποίηση τη μα Κυρία και έχει ο κύριο Ροσφόρ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Βασικά έχω αναρρύθμιτες ερωτήσει γιατί είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να τις ταξινομήσω λίγο και να μην θέσω κάποιε από αυτές τι ερωτήσεις. Λοιπόν, από όλε τι παρεμβάσει των εμπειρογνωμόνων άκουσα Πώ θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από αυτέ τι πρόταση, παρότι βέβαια η εκτίμησή του από την πλευρά του, ε, εκτίμηση τη πρόταση ήταν διαφορετική. Και επίση άκουσα με κάποια συνοχή, ε, όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά από όλου, ότι ε, θα πρέπει να έχουμε μια κάπω μεικτή προσέγγιση όπου αυτό χρειάζεται, ενώ σε άλλε περιπτώσει, σε άλλου τομεί θα πρέπει να κινηθούμε προ την κατεύθυνση τη ελάχιστη εναρμόνισης αυτό φανταζόμουν και εγώ και το βλέπω τώρα να επιβεβαιώνεται εκ νέου. Έχω ε, να θέσω ένα δύο συγκεκριμένα ερωτήματα στον κύριο Σανασό από την Φόρμπερκ. Μας δώσατε λοιπόν κάποια πολύ όμορφα παραδείγματα, αλλά εξετάζοντας αυτά τα παραδείγματα είδα ότι είναι πάρα πολύ επιλεκτικά και στα οποία βέβαια έχει τονιστεί με ιδιαίτερο τρόπο οτιδήποτε πιο θετικό. Όμως, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη σελίδα 8 της δικής σας ε, παρουσίασης, ε, όπου αναφέρεστε ε, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, λέτε ας πούμε σε σύναψη του Συμβουλίου 9 Οκτωβρίου και μετά παναχώρηση. Εάν δεν περιλαμβάναμε αυτό το στοιχείο εδώ, πώς θα διαμορφώνονταν χρωματικά αυτός ο χάρτης εδώ, δεν θα αναζάλλει τελείως τα πράγματα. Νομίζω πως είναι επικίνδυνο για όλους τόσο δηλαδή για αυτού που είναι υπέρ, όσο και για αυτού που είναι κατά, να βασιζόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα, γιατί κάτι τέτοιο δεν απηχεί το πνεύμα τη ε, νομοθετική πρόταση. Ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό ήταν μια παρατήρηση. Τώρα θα ήθελα να θέσω το ερώτημα αυτό καθε αυτό. Εσείς ως εκπρόσωπος εδώ αυτής της Φόρβερκ ε, και της ε, Forver και ε, πήγα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και εξέτασα την ιστοσελίδα σας, είδα τα προϊόντα σας, δεν υπάρχει κάτι λανθασμένο. Πήγα όμως στο forwerk.de, forwerk.fr και forwerk.be, δηλαδή Γερμανίας, Γαλλίας, Βελγίου τα site και είδα πολύ διαφορετικές σελίδες στις οποίες είχαμε πολύ διαφορετικά προϊόντα τα οποία ε, διαθέτουν οι δικές σας επιχειρήσεις και δεν είδα σε καμία από αυτές τις ιστοσελίδες ε, τιμοκατάλογο τελικά των προϊόντων. Είτε λοιπόν αυτός ο τιμοκατάλογος δεν υπήρχε καθόλου, είτε είναι κάπου κρυμμένος εκεί μέσα, πολύ καλά κρυμμένος. Άρα λοιπόν, το ερώτημά μου, αφού έχετε τρεις πολύ διαφορετικές ιστοσελίδες, στις οποίες ε, και εν μέρει διαφορετικά προϊόντα, ένα γεγονός το οποίο δεν σχετίζεται τόσο με την νομοθεσία αλλά με τις ε, ανάγκες τελικά των καταναλωτών. Δηλαδή σκέφτεσαι το τι μπορεί κανείς να πουλήσει πού. Άρα λοιπόν σας ζητώ να μου διευκρινίσετε ότι ακόμα και αν προβαίναμε σε μια πλήρη εναρμόνιση όλων αυτών των σημείων τα οποία θεωρείται σωστά, θα, θα ανοίγαμε την ιστοσελίδα σας και θα είχαμε μια ενιαία ιστοσελίδα και δεν θα προσφέρονταν ε, διαφορετικά προϊόντα. Λαμβανομένου υπόψη σας λέω ότι τελικά οι ανάγκες των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα είναι διαφορετικές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ευχαριστώ για την ερώτηση και επειδή είχατε διαβάσει καλά το μάθημά σας. Ο κύριος Ροσφόρ και μετά θα ακούσουμε κάποιες απαντήσεις. κύριος Ροσφόρ, θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Business Europe αν τα όσα είπε είναι όντως αντιπροσωπευτικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι μόνο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Γιατί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνήθως έχουν μία αγορά πολύ τοπική, πολύ εθνική. Μήπως λοιπόν θα αντιμετωπίσουν κίνδυνο αποστεθεροποίησης εξαιτίας ε, της αποδιάρθρωσης του εθνικού νόμου, της εθνικής νομοθεσίας. Και μία ερώτηση προς την κυρία Γκογιάνς θεωρώ ότι από πλευράς προστασίας καταναλωτή κάτι που πρέπει να λέμε συναχώς είναι ότι σήμερα όπου και να ζει κανείς ο καταναλωτής δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του. Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της οδηγίας είναι ότι από τη στιγμή που έστω και σε ένα πεδίο θα υπάρξει εναρμόνιση έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε σε μεγάλη κλίμακα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους. Αυτό νομίζω ότι είναι θεμελιώδους σημασίας, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι αντιφατικό να αναπτύσσουμε παράλληλα την εσωτερική αγορά και τις επιχειρήσεις και την προστασία του καταναλωτή. Γιατί πάντα ο καλύτερος καταναλωτής οπουδήποτε στον κόσμο και άρα και στην Ευρώπη είναι ο καταναλωτής που γνωρίζει τα δικαιώματά του. Και μετά από αυτό που εκεί είπε και η κυρία Γκέπχαρτ, όντως χρειαζόμαστε πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν και αναρωτιέμαι αν για ένα τόσο πολύπλοκο θέμα θα καταλήξουμε κάποια στιγμή να έχουμε μια ανάλυση αντικτύπου που θα καλύπτει τα πάντα, ακόμη και το ψυχολογικό αντίκτυπο, αν θέλετε, για τους καταναλωτές. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε έναν καλό συμβιβαστό συμβιβασμό μέσω της μεικτής εναρμόνισης. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η Κομισιόν με μια τέτοια προσέγγιση. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική της άποψη. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρόσφορ και κυρία Ρούλερ. Είχα ζητήσει το λόγο πρωτού πάρει το λόγο η κυρία Γκέμπχαρτ, ο κύριος Σφάμπ και η κυρία Γκέμπχαρτ ε, κάλυψε ε, σε μεγάλο βαθμό ότι αυτό δυστυχώ θα πρέπει να συνταμίσω πάρα πολύ. Ε, πράγματι θεωρώ πω χρειαζόμαστε εδώ μια μεικτή προσέγγιση. Υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εναρμονιστούν και μάλιστα ε, και πλήρω και θα πρέπει να βρούμε μια λύση, αλλά από την άλλη πλευρά ε, δημιουργεί και πολλέ ασάφειε, περισσότερε ασάφειε παρά βεβαιότητε με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι σε αυτό που ανέφερε η κυρία Γκέπχαρτ. Δηλαδή, οι μεγάλε επιχειρήσει οι οποίε έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν το πώ διαμορφώνεται η κατάσταση για αυτέ τι διάφορε ε, ε, χώρε, στα 27 κράτη-μέλη, δεν έχουν πρόβλημα. Μπορούν δηλαδή να προβούν και σε μελέτε σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά των καταναλωτών και στο στοχοθετούν, εστιάζουν δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένε ηλικιακέ ομάδε ε, και ούτω καθεξή, γιατί γνωρίζουν πω ε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο τα ίδια κράτη-μέλη. Έχουν δηλαδή διαφορετική ε, αγοραστική συμπεριφορά, διαφορετικέ πολιτισμικέ παραστάσει οι πολίτε και οι κατανότε των διαφορών κρατών μελών. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω για μία ακόμα φορά. Αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε πω θα αποτελούσε πρόοδο μία μεικτή εναρμόνιση και νομίζω πως ο εκπρόσωπος της Φόρτβεκ θα συμφωνούσε με αυτό. Είχαμε και μια εκ των προτένων συζήτηση, είχατε πει πως ε, με κάποιες ε, διευκολύνσεις στο τεχνικό τομέα πολλά θα μπορούσαμε να επιτύχουμε, αλλά ε, το δεύτερο τμήμα της πρότασης σας δεν είναι και τόσο σοβαρό. Ευχαριστώ. Right. Άλλοι συνάδελφοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν ε, περίπου ίσες ερωτήσεις για όλους. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τις απαντήσεις και ελπίζω να καταλάβετε αν απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματά σας. Ο κύριος Αλβάρας, ευχαριστώ. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θεωρώ ότι οι βασικοί που θα ωφεληθούν είναι ακριβώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν αυτή τη στιγμή να διαφοροποιούν την πρακτική τους ανάλογα με το κάθε κράτος και τις διατάξεις του. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να πολλούν τα προϊόντα τους εκτός της επικράτειας του κράτους τους. Γι' αυτό λοιπόν από πλευράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων στηρίζουμε αυτή την νομοθεσία και να πω ότι η δική μας οργάνωση εκπροσωπεί σαφώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ένα σχόλιο για την πλήρη εναρμόνιση και το σχόλιο του κυρίου Σμιτ για τις επιχειρηματικές οργανώσεις είναι σαφές ότι ο βασικός στόχος και το βασικό όφελος αυτής της πρότασης είναι, ένα πλήρη, μια πλήρης εναρμόνιση. Δεν θέλουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση, γιατί αυτό πάλι θα οδηγήσει σε 27 διαφορετικές μορφές και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Δεν ξέρω πόσο μεγάλες θα είναι οι αλλαγές, όμως η πλήρης εναρμόνιση θα ωφελήσει και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που θα έχουν τα ίδια δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω καταρχάς στην κυρία Γκέμχαρτ. Σας ευχαριστώ για, την, ε, ένδια, για το ενδιαφέρον σας ε, για την εταιρεία μας. Δεν ξέρω σε ποιο site μπήκατε. Όμως έχουμε μία περιορισμένη σειρά προϊόντων και πολλούμε όλα τα προϊόντα σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε διάφορες θηγατρικές σε 11 διαφορετικά κράτη-μέλη, πράγμα λογικό εφόσον δραστηριοποιούμαστε τα τελευταία 126 χρόνια. Και ιστορικά προσπαθούσαμε πάντα να δημιουργούμε διαφορετικές θηγατρικές στα κράτη-μέλη αντί να κάνουμε διασυνοριακές πωλήσει. Πάντως, αυτές ε, οι 11 θηγατρικές δραστηριοποιούνται συνολικά σε 23 κράτη-μέλη. Βρήκατε λοιπόν τη γαλλική, τη Βέλγια και τη γερμανική θηγατρική μας που πολλούν τα ίδια προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους. Βεβαίως, μπορούμε εδώ να παίξουμε με ερωμηνίε ή με οτιδήποτε άλλο, αλλά η πραγματικότητα, αυτό που έχει σημασία, δεν είναι η μία παράβρετρος που βρήκατε εκεί για το δικαίωμα απόρριψης. Δεν έχει να κάνει με την ονομαστική προθεσμία, αλλά με την πραγματική προθεσμία αν λάβουμε όλους τους κανόνες υπόψης τους κανόνες που αφορούν ε, την πληροφόρηση, τη λήξη κτλ. κτλ. Για παράδειγμα, να σας δείξω πώς ε, αυξάνεται παντού η προστασία των καταναλωτών. Άμα το ψάξω μπορώ να σας βρω ένα παράδειγμα για κάτι που συμβαίνει αυτό και βελτιώνονται παντού τα πράγματα, όπως μπορώ να σας βρω και παράδειγμα για το αντίθετο. Τώρα, για να απαντήσω στην κυρία Ρούλε. Αμφιβάλλεται για τις εγγύησει και για αυτά που είπα σχετικά με τις εγγύησει. Λυπάμαι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε το λανθασμένο στην παρουσίασή μου. Παρακαλώ, Διαβάστε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει, της Eurocommerce, της Business Europe, του κυρίου Σούλτνερ, του Legal Compendium, όλες τις μελέτες. Ναι, θα μπορούσα να είχα χρησιμοποιήσει άλλα παραδείγματα. Πάλι παρόμοια όμως θα ήταν. Για τα βασικά κριτήρια, δικαίωμα υπαναχώρησης, προθεσμία, καθώς και αντιστροφή του βάρους απόδειξης, τελικά ναι, υπάρχουν, υπάρχει μία μείωση της προστασίας σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά συνολικά αυξάνεται η προστασία. Και αυτό είναι σαφές. Να απαντήσω στην τελευταία απάντηση. Ναι, αν δείτε μόνο την εφαρμογή της οδηγίας ισχύει αυτό, αλλά άμα δούμε το σύνολο της αστικής νομοθεσίας σε κάθε κράτος μέλος, για αυτό το σύνολο ο πίνακας δεν ισχύει πλέον, είναι απαρχαιωμένος. Και θα ήθελα να πω και στον κύριο Σφάμπα ότι όταν μιλάμε για ελάχιστη εναρμόνιση θεωρήθηκε ότι η ελάχιστη εναρμόνιση ήταν νίκη για τα δικαιώματα του καταναλωτή και μπήκε και στη συνθήκη του Μάστρεχτ. Οπότε, τα τελευταία χρόνια έχουμε προσπαθήσει πολύ για να μην είμαστε δογματικοί, αλλά ρεαλιστές. Και αυτό το έχουμε κάνει σε συνεργασία με όλες τις οργανώσεις μέλη μας. Και γι' αυτό λέμε για αυτή την πρόταση ότι μπορούμε να δεχτούμε μία μεικτή προσέγγιση με πλήρη εναρμόνιση για τα τεχνικά θέματα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν διασυνοριακές πωλήσει, όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτε άλλο εκτός από στην ελάχιστη ενημέρωση όσον αφορά τις νομικές εγγύησεις. Και λυπόμαστε πολύ γιατί η κυρία Κουνέβα μας λέει ότι δεν μπορεί να δεχτεί οτιδήποτε άλλο εκτός από πλήρη εναρμόνιση. Γιατί νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Και να απαντήσω στον κύριο Ροσφόρ. Όταν ε, εργάζεστε για ένα κίνημα καταναλωτών πρέπει να θυμάστε ότι δεν υπάρχει μόνο ένα βήμα. Σίγουρα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής τα δικαιώματά του και η οργάνωση θα προσπαθήσει να κάνει μία εκστρατεία ενημέρωσης, είτε αυτή είναι ευρωπαϊκή, είτε εθνική, είτε κρατική, είτε προέρχεται από τις οργανώσεις των καταναλωτών. Και μετά πρέπει να έχουμε και την εφαρμογή της νομοθεσίας, δηλαδή διαχείριση των προσφυγών, διακανονισμοί, Αν και θεωρώ ότι αυτό το θέμα δεν είναι το θέμα της σημερινής ακρόασης, παρόλο που για εμάς και αυτός ο τρίτος πυλώνας είναι πολύ σημαντικός. Δεν δέχτηκα ερωτήματα εγώ, αλλά θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Ροσφόρ. Ναι, όπως είπε και η Μονίκ, έχουμε πρόοδο κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν κάποια θέματα όπως ο Ευρωπαϊκός Οδηγός για το ηλεκτρονικό εμπόριο που μας δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια ελάχιστη προστασία. Όμως, ακόμα και αν πετύχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση, υπάρχει κάτι που παραμένει. Τι οι νομικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Εκεί τι γίνεται έχει δικαίωμα λύση της σύμβασης ε, ο καταναλωτής κτλ. Αυτό το θέμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών αυτή τη στιγμή και περιλαμβάνει διάφορες νομικές πτυχές. Και εκεί παίζεται το παιχνίδι, όμως αυτή η πτυχή είναι κάτι που μας διαφέρει αυτή τη στιγμή. Οπότε ζητάμε από την Κομισιόν να σταματήσει να χρησιμοποιεί το σύνθημα της πλήρους εναρμόνισης γιατί εφόσον υπάρχει αυτή η νομική πληρονομή, πλη, ποικιλομορφία μας συγχωρείτε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή την ποικιλομορφία. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τώρα, αν κάποια στιγμή γίνει αυτό που έγινε και με την οδηγία για την πίστοση. Ναι, από τη μία πλευρά μιλάμε για πλήρη εναρμόνιση και εκεί, από την άλλη κάποιες αρμοδιότητες παραμένουν στα κράτη-μέλη. Οπότε, στα πιο ευαίσθητα σημεία χρειάζεται να υπάρξει μία ελάχιστη εναρμόνιση. Γιατί ναι, μεν μπορεί να θέλουμε όλοι να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε και να πέσουμε πάνω στον τοίχο. Ναι, πάντως η οδηγία για τους καταναλωτές προσπάθησε να έχει εναρμόνιση. Αυτή ήταν και η ορολογία που χρησιμοποιήσαμε. και δεν ξέρω αν ε, είχαμε αλλάξει κάτι, αν θα μας είχε βοηθήσει στην έγκριση. Εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα ενδιαφέροντα και συμπληρωματικά στοιχεία που μας δώσατε, καθώς και για τη σαφήνεια των λόγων σας. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντόιλινγκ από την πλευρά της Προεδρίας του Συμβουλίου και μετά στην κυρία Τεστόρη από πλευράς Επιτροπής. Μετά θα δούμε αν υπάρχουν άλλα αναπάντητα ερωτήματα από τους συναδέλφους και τέλος θα δώσω το λόγο στην εισηγητή ο οποίος θα προσπαθήσει να συνοψίσει τα πάντα. Αν και αυτό θα πρέπει να είναι πραγματικά αριστούργημα και πολύ δύσκολο έργο για να το καταφέρει. Αλλά τον βλέπω που κρατάει σημειώσεις. Οπότε, αν δεν κάνω λάθος, δεν είστε ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας. Παρ' όλα αυτά, εκπροσωπείτε τη Σουηδική Προεδρία. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μας καλέσατε σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η νομοθεσία για τη Σουηδική Προεδρία και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την επίτευξη προέδρου, προόδου. Ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ σήμερα και ακούμε τις συζητήσει αυτές, ιδιαίτερα παραγωγικές και ενδιαφέρουσες. Η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της πέρυσι τον Οκτώβριο και οι συζητήσεις στο Συμβούλιο ξεκίνησαν επί Γαλλικής Προεδρίας, στο τέλος της Γαλλικής Προεδρίας που διοργάνωσε και μία συνδιάσκεψη με κύριο θέμα ε, την ε, οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Στη συνέχεια, η Τσεχική Προεδρία ε, οργάνωσε τακτικέ ε, συναντήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε ερωτήσεις προ την Επιτροπή, να δούμε ορισμένα προβλήματα τα οποία ε, προέκυψαν. Με δύο λόγια, δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουν τα θέματα αυτά τα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι ε, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια μπορέσαμε να αποκρισταλώσουμε τις απόψεις και τους τομεί που παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πού χρειαζόμαστε περισσότερη προσέγγιση, αν θέλετε. Και στην 1η Ιουλίου που ανέλαβε ε, η Σουηδία την Προεδρία, αναλάβαμε, πήραμε τη σκητάλη για το θέμα αυτό, συνεχίσαμε τις τακτικές αυτές συνεδριάσεις, ξεκινήσαμε εξετάζοντα το κεφάλαιο 4 που αφορά τα λαθηματικά προϊόντα και στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τη γενική συζήτηση για, τις, για τους αυθέμητους ε, ε, συμβατικούς όρους. Δεν έχουμε εξετάσει όμως ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει την εξέταση των θεμάτων αυτών. Γιατί υπάρχουν διάφοροι εθνικοί κατάλογοι και πρέπει να δούμε πώς, θα συνδε... πώς, παραπέμπουμε στους καταλόγους αυτούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα ε, ε, που εργάζεται επί του θέματος αυτού στη Στοκχόλμη για να δούμε πώς μπορούμε να το προωθήσουμε και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το πεδίο εφαρμογής. Στόχος είναι να δούμε όλες τις πτυχές της οδηγίας ε, επί Σουηδικής Προεδρίας. Η εντύπωσή μας ε, είναι ότι οι συζητήσει είναι επικοδομητικέ και χρήσιμε στο Συμβούλιο. Πάντω είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε το γεγονό ότι απέχουμε ακόμα πολύ από οποιαδήποτε ε, συμφωνία πραγματική συμφωνία ή ε, συνένεση σε κάποιο τομέα. Αλλά όλοι έχουμε την εντύπωση ότι όλοι οδεύουν προ την ίδια κατεύθυνση, σωστή κατεύθυνση. Και τα κράτη-μέλη καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να μπορέσουν να προτείνουν συγκεκριμένε λύσει στα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν. Νομίζω ότι τα ερωτήματα τα οποία ε, ήταν ε, τα πιο αμφιλεγόμενα και τα οποία συζητήθηκαν περισσότερο στα κράτη-μέλη αφορούν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας το συζητήσαμε σήμερα. Μιλήσαμε για το νησί και τη θάλασσα, το νησί και τον ωκεανό. Ε, να προσπαθήσουμε λοιπόν να προσδιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή. Ναι, όσον αφορά αυτό το μέτωπο, χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια ε, στο κείμενο τη οδηγία. Και στη συνέχεια έχουμε το θέμα των σχέσεων, τις σχέσεις με το δικαίωμα σύναψη συμφωνίας και με ε, την νομοθεσία συνολικά ε, για τι συμφωνίε και τι συμβάσει και το πώ όλα αυτά ε, θίγονται από, και επηρεάζονται από την παρούσα πρόταση. Τώρα, θα τα επεξεργαστούμε όλα αυτά μέσα στο φθινόπωρο και στι αρχέ ε, Δεκεμβρίου έχουμε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα. που Εκεί οι Υπουργοί για θέματα κατανάλωση θα συζητήσουν ε, τα θέματα με του ομολόγου του ε, των άλλων κρατομελών. Είναι δύσκολο να δούμε από τώρα μέχρι ποιο σημείο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα, στο χρονικό περιθώριο που έχουμε και τι θα μπορέσουμε να έχουμε πετύχει. Πάντω σίγουρα ελπίζουμε να σημειώσουμε ώστε εδώ περισσότερη πρόοδο. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το σχέδιο οδηγία Και όσον αφορά τα σχόλια της Υπουργού για θέματα κατανάλωσης, όταν ήρθε εδώ είπε ότι η Σουηδική Προεδρία με μεγάλη χαρά περιμένει τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας και ε, ε, είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε την παραμικρή συνδρομή. Αυτά θέλω να πω και σε ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω, αν μου επιτρέπετε, να σας κάνω ένα ερώτημα. Γιατί νομίζω ότι έχει σχέση με τη συζήτηση που είχαμε. Ίσως λοιπόν μπορείτε να με διαφωτίσετε. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει στόχο ε, την κατεύθυνση ε, της μέγιστης ε, εναρμόνισης ή θα μπορούσαν να υπάρχουν κάτι μέλη που μπορούσαν να δεχτούν μια μεικτή προσέγγιση ε, όπως αυτή την οποία ανέφερε η κυρία Γκόγεμς ή βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις μας αφορούν την ουσία της πρότασης Δηλαδή στηριζόμαστε την πρόταση της Επιτροπής. Δεν, ε, δεν κάνουμε συγκεκριμένε συζητήσει για την εναρμόνιση. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τα θέματα κεφάλαιο προ κεφάλαιο και βλέπουμε πώ μπορούμε να βρούμε λύσει και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Εξετάζουμε λοιπόν την πρόταση, που βεβαίω ο τελικό στόχο τη είναι η πλήρη εναρμόνιση. Αλλά τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα εξετάσει το άρθρο 4 που αναφέρεται στο επίπεδο εναρμόνιση αναφερθήκαμε στην ουσία τη ε, οδηγία, στο σύνολό τη και δεν ασχοληθήκαμε με την εναρμόνιση. Πολύ αποκαλυπτική απάντησή σα. Ευχαριστώ. Όχι. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα ε, την πρόσωπο της Επιτροπής που κάθισε ε, όλο το απόγευμα και κράτησε και σημειώσεις. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε, κύριε Τεστόρη. Ίσως λοιπόν θέλετε να μας δώσετε την εντύπωσή σας μέχρι στιγμής. Και αν έχετε κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι η μεγάλη τιμή για μένα ε, που μου δίνετε λίγα λεπτά για να απαντήσω εμείς είμαστε η υπηρεσία υπεύθυνη για θέματα καταναλωτών. Αυτό που θέλουμε είναι να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις δυνατότητες επιλογής τους. Η πρότασή μας έγινε πριν από ένα χρόνο και όπως σας είπα, όπως είπε και η Επίτροπος, είμαστε έτοιμοι να βελτιώσουμε τα πράγματα και να ξαναδούμε το επίπεδο προστασίας. Ήδη σας ανέφερα ε, τις εγγυήσεις στα ένδικα μέσα. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μας και στο Συμβούλιο και, και συζητήσει με το Συμβούλιο. Πρέπει να σα πω το εξή: Μίλησα για ένα νησί πλήρη εναρμόνιση σημαίνει πλήρη εναρμόνιση του νησιού και όχι ολόκληρη τη θάλασσα. Υπάρχουν τομεί που δεν εναρμονίζουμε. Ε, ε, ε ικανότητα ε, για σύμβαση, υποχρεώσει, ευθύνε. Δεν εναρμονίζουμε τα πάντα. Δικαιοπραξία. Εμεί ασχολούμαστε με ορισμένα συγκεκριμένα σημεία και δεν ασχολούμαστε, ασχολούμαστε με το σύνολο. I would like to answer, you know, to... Και να σα πω και κάτι άλλο. και απευθύνομαι στη Μονίκ ε, γιατί μερικές φορές διαφωνούμε. Ποια, ποια είναι τα πραγματικά εμπόδια για περισσότερες διασυνοριακές συναλλαγές. Γιατί οι περισσότερε διασυνοριακέ συναλλαγέ αποτελούν προστιθόμενη αξία για την οικονομική ανάπτυξη. Δεν νομίζω ότι κανεί διαφωνεί, ούτε κι εσεί. Όχι μόνο λοιπόν αποτελεί ένα πλεονέκτημα για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για τον καταναλωτή, γιατί έχει περισσότερε επιλογέ. Και ειλικρινά, θέλω να σα καλέσω να διαβάσετε, γιατί εμεί, μα πήρε 9 μήνε η αξιολόγηση αντικτύπου εκφράζουμε αριθμητικά το κόστος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα του κόστους. Για ε, τις πωλήσει εξ αποστάσεως. 30 φορές λιγότερο θα κοστίζει ε, η πώληση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι για, την για το κατακαιρματισμό, αλλά υπάρχει ο κατακαιρματισμός. Και ακριβώς για αυτό το λόγο η παράδοση είναι πιο περίπλοκη. Το πρόβλημα της γλώσσας είναι ε, ε, διαφορετικό. Ευτυχώς έχουμε 22 διαφορετικές γλώσσες και κανείς δεν θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Και κάτι άλλο. Όχι, κοιτάξτε, ειλικρινά σας το λέω όταν λέμε ότι ο πίνακά μα δεν είναι πλήρη, δεν είναι καλό, ε, δεν είναι ε, σαφή. Εντάξει, σωστά είναι όλα αυτά. Αλλά ε, πρόκειται για συνεχιζόμενη εργασία. Εμεί θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σα με πλήρη διαφάνεια κάτι που δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο τη Επιτροπή. Ακριβώ αυτό το λέμε ανεπίσημο έγγραφο, non-paper. Δεν μπορούμε αυτό το χρονικό διάστημα να έχουμε επίσημο έγγραφο τη Επιτροπή. Θα υπάρξει όταν θα υπάρξουν τροπολογίε και θα πάρουμε θέση. Άρα ε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε ένα ε, διαφανή και ανοιχτό διάλογο με όλους σας και με όλους τους ενδιαφερόμενους. Ευχαριστώ. Uh, well, ladies and gentlemen. Ε, τις 6, ε, έχουμε και το χρόνο ακόμα, αλλά πρωτού ζητήσω από τον ε, Αντρέα Σόμπ να συνοψίσει τη συζήτηση. Εάν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να πάρει το λόγο, ναι, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία, αφού έχουμε αυτή την, αυτό τον περισσότερο χρόνο και αφού βρίσκονται εδώ οι εμπειρογνώμονες μαζί μας. Ε, θα ήθελα ε, να πω κάτι στην κυρία Τεστόρη. Ε, μόλις τώρα μας είπε ότι επιθυμεί ε, μόνο πλήρη εναρμόνιση του νησιού, όχι όλη τη θάλασσα. Η κυρία Κούνεβα όμω, ε, όταν τη ρωτήσαμε σχετικά, μα έδωσε μια τελείω διαφορετική εντύπωση. Είπε πω δεν ε, πρόκειται κανένα να την αποτρέψει από το στόχο τη να επιτύχει πλήρη εναρμόνιση σε αυτό το τομέα. Προφανώς μπορούμε να ασχοληθούμε με ζητήματα ορισμού του αντικειμένου με το οποίο ασχολούμαστε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει διευκρινίστε λίγο τη, τη, τη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί θέλετε να μιλήσετε τελικά. Δεύτερο ε, ζήτημα που θα ήθελα να αναφέρω. Και εδώ και πάλι απευθύνομαι στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επανέρχομαι σε ένα ζήτημα το οποίο είχαμε κατά την πρώτη ακρόαση και ένα ερώτημα το οποίο είχε θέσει ο κύριο ε, Σφαμπ. Πολύ ενδιαφέρον ε, ερώτημα. Ήταν ένα εμπειρογνώμονα, εδώ νομικό εμπειρογνώμονα, δεν έχω ξεχάσει το όνομα. Αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Και μα είχε δείξει λοιπόν αυτή η εμπειρογνώμονα ε, μια σύγκριση μεταξύ, διο, μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, με του Κιέλου και του Σασβούργου όπου έχουμε δύο αγοραστέ οι οποίοι έρχονται, προβαίνουν σε μια, στη σύναψη μια συμφωνία για ένα ε, εργαλείο το οποίο επιθυμούν να αγοράσουν και στη συνέχεια αποφασίσουν να επαναχωρήσουν από αυτό το συμβόλαιο. Και ε, κάποιο ε, από, την Γαλλία αναρωτιέται πώ γίνεται δυνατόν αυτό να μην ισχύει στη Γερμανία. Ε, κύριε Σουάμπ, Εσεί είχατε πει πως το δίκαιο σε αυτέ τι δύο διαφορετικέ χώρε είναι διαφορετικό. Ότι υπάρχουν δηλαδή κάποια δικά δικαιώματα στο γαλλικό δίκαιο τα οποία δεν ισχύουν στο γερμανικό. Η εμπειρογνώμονα ε, νομικό μα είπε πω όχι. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Το δίκαιο στι δύο αυτές χώρε είναι το ίδιο. Όμω οι συνέπειε, τελικά του ίδιου αυτού δικαίου είναι διαφορετικέ. Διαφορετικές γιατί ε, στην ε, Γαλλία υπάρχει διαφορετική διαμόρφωση του από Υπάρχει δηλαδή το διαφορετικό δικαίωμα Κούλιγκοφ στη Γαλλία από ότι στη Γερμανία. Δηλαδή είναι πιο εύκολο τελικά για ένα καταναλωτή να υπαναχωρήσει από αυτή τη σύμβαση. Υπάρχει δηλαδή διαφορετική εφαρμογή ίδιας νομοθεσίας. Και αυτό ήταν το ζήτημα για μένα. Και αυτό είναι το ερώτημά μου στην εκπρόσωπο, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιου είδους πολιτισμικές εντός εισαγωγικών διαφορές και μπορούν να επιληθούν αυτέ μέσω μια τέτοια πρόταση. Εγώ νομίζω πω δεν μπορούμε να το επιτύχουμε. Και νομίζω πως ε, ο κύριος ε, Σμίτς ε, καταλαβαίνω από νεύμα του ότι δεν συμφωνεί μαζί μου. Μάλλον κάνω κάποιο λάθο, δεν ξέρω. Α μου διευκρινίσει ποιο είναι το λάθο μου. Απευθύνομαι λοιπόν και στον κύριο Σμιτ. Γιατί ε, πρόκειται για ένα πεδίο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε οπωσδήποτε υπόψη στη συζήτησή μας. Πολλοί εμπειρογνώμονες και εμπειρογνώμονες τώρα μίλησαν πολύ για την αγορά, μίλησαν πολύ για το δίκαιο, αλλά δεν μίλησαν πολύ για τους καταναλωτές. Ε, για δεύτερη φορά λοιπόν κάνω την απόπειρα σήμερα να κατευθύνω τη συζήτηση προς τους ίδιους τους καταναλωτές, πράγμα το οποίο δεν κατάφερα μέχρι στιγμής. Ελπίζω να το καταφέρω τώρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ έχω την κυρία την κυρία Στάιλερ, κάποιος άλλος από την Επιτροπή που θέλει να κάνει κάποια τελευταία ερώτηση. Η κυρία Σαρτεμόζα. Er Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. όπω είπε και η Εύελιν και εγώ θεωρώ ότι επειδή έχουμε λίγο χρόνο, α τον αξιοποιήσουμε ώστε να τον καλύτερα. Γι' αυτό πήρε το λόγο. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα υπόθηκαν σήμερα εδώ σε αυτήν την Πρέπει να σα πω ότι το σκέφτηκα το ζήτημα. Και είναι μπερδεμένη γιατί μερικέ φορέ έχω την εντύπωση ότι συζητάμε άλλη πρόταση. Ακούω την Επιτροπή και ακούω και του εκπροσώπου των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και έχω την εντύπωση ότι για άλλο μιλάει ο καθένα. Άρα λοιπόν οι απόψει δίστανται ιδιαίτερα. Ποιο, ε, για να δούμε τώρα, ποιο είναι το, κεντρικό σημείο τη συζήτηση σήμερα. Ότι Εντάξει, υπάρχουν αυτέ τι διαφορέ, γιατί έχουμε διαφορετικέ προοπτικέ και διαφορετικέ οπτικέ γωνίε όταν συζητάμε τα ζητήματα αυτά. Και υπάρχουν αυτέ τι διαφορέ στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πλήρη εναρμόνιση είναι υπέρ των επιχειρήσεων. Αλλά από την άλλη, έχουμε κάποιε επιφυλάξει. Γιατί αν εξετάσουμε το θέμα από τη σκοπιά του πολίτη, του καταναλωτή, και προσπαθούμε να δούμε τα πλεονεκτήματα, μα δεν μπορούμε να τα δούμε τουλάχιστον άμεσα. Τώρα η Επιτροπή μας λέει ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής, όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα ε, ωφεληθούν από την πρόταση. Εντάξει, ωραία. Αλλά ίσως ήταν καλύτερο η Επιτροπή να μας πει ότι παρουσιάζουμε την πρόταση αυτή γιατί θέλουμε να προωθήσουμε το διασυνοριακό εμπόριο και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Στη χώρα μου, στη Δανία, στις ευρωεκλογέ αυτό ε, το ζήτημα ήταν ένα βασικό ζήτημα. Από τη μια μεριά δηλαδή η προστασία των καταναλωτών και από την άλλη η, εναρμόνιση ή μη μια σειρά κανόνων από τις Βρυξέλλες. Άρα λοιπόν ο, ο πολίτης πρέπει να μπορεί να δει τα πλεονεκτήματα μιας, ε, της πρότασης. Γιατί αν δεν μπορεί να τα δει τότε έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να εξετάσουμε σε όλες τι λεπτομέρειε ε, την πρόταση και να δούμε ποιε θα είναι οι επιπτώσει. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το βαλάκι είναι πάλι από τη μεριά της Επιτροπής. Η κατάσταση ε, διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, αλλά ο πίνακα ε, που επεξεργάστηκε η Επιτροπή Ακριβώ για αυτό το σκοπό δεν μπορεί να είναι, για αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι διεξοδικό. 27 κοινοβούλια. 27 εθνικά κοινοβούλια. Ε, κοιτάξτε, ίσω θα πρέπει να ζητήσουμε την άποψή του απευθεία, να του αποστείλουμε μια επιστολή και να μα πούνε τι πιστεύουν, να ε, ε, ακούσουμε και την άποψή του. Δεν αρκεί η αξιολόγηση τη Επιτροπή. Σίγουρα η πρόταση της Επιτροπής ε, θα βοηθήσει τις, ε, τις επιχειρήσεις, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μάθω τι πιστεύω και τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί με ενδιαφέρει η πρόταση να μην είναι μόνο προς όφελος των επιχειρήσεων, αλλά και των καταναλωτών. Ε, ε πρόεδρος. Μα είχαμε ήδη μία συνεδρίαση και μία συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για το ζήτημα αυτό. Ίσως όμως ο εισηγητή να σκεφτεί ε, ότι θα έπρεπε να γίνει και άλλη μία συνάντηση. Θα έπρεπε ίσως να ακούσουμε την άποψη των Εθνικών Κοινοβουλίων για άλλη μια φορά. Κύριε Στάιλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές σε σχέση με αυτά που είπε η Εύελιν και η Κρίστα. Να σα πω το εξή. Σίγουρα στη δική μου εκλογική περιφέρεια, στη Σκωτία και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν φόβοι σε σχέση με τη μείωση προστασία των καταναλωτών, ε, ελαττωματικά αγαθά για παράδειγμα, ε, δικαίωμα ε, λύση τη σύμβαση. Κοιτάξτε, όλα αυτά και βλέπω στην πρώτη επιτροπή, δεν νομίζω ότι ενισχύονται τα, τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κοιτάξτε, σε αυτέ τι διαφάνειε, σε αυτή την ενημέρωση, σελίδα 12, υπάρχει ένας πολύ χρήσιμο πίνακας Και βλέπω και μια σκοτσέζικη σημαία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, αυτό δείχνει ακριβώς ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και Σκοτία συγκεκριμένα θα, μειωθούν, ε, θα, μειωθεί μειωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών με βάση το άρθρο 20 για, ε, για την ε, διετή εγγύηση. Μα εκεί θα έχουμε μείωση της προστασίας των καταναλωτών και όχι αύξηση. Στην σελίδα 13 επίσης Εκεί βλέπουμε πάλι το πώς θα επηρεαστούν όλα τα κράτη-μέλη. Και σε 12. Άρα το ερώτημα παραμένει. Σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα πώ μπορούμε να μιλήσουμε για ενίσχυση, πώ εγώ θα πω στου ανθρώπου που εκπροσωπώ ότι ενισχύεται η προστασία του, όταν μειώνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει τόσα πολλά, τόσα πολλά σημεία που πρέπει να εξετάσουμε στι ε, λεπτομέρειέ του. Και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα σήμερα το απόγευμα, αλλά πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και βέβαια έχω κι εγώ πολύ υλικό για σκέψη. Και ζω και σε ένα νησί, οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να το σκεφτώ το θέμα πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ, Κάθριν. Να σα ρωτήσω ε, το εξή. Στην ίδια σελίδα. υπάρχει πρόβλημα με το διασυναριακό εμπόριο ανάμεσα στη Σκωτία και στην Αγγλία. Γιατί έχετε διαφορετικές ε, ε, περιόδους ευθύνης. Α, θα αυτό το θέμα, θα το συζητήσω και με την ε, κυβέρνηση της Σκωτίας. Δεν θέλετε εκεί πέρα να έχετε ελάχιστη εναρμόνιση. Ωραία. Ε, ε, είχαμε αρκετές ερωτήσεις. Να δώσουμε λοιπόν την κυρία Τεστόρη το λόγο για να έχει την τελευταία λέξη. Νομίζω όμως ότι υπήρξαν και ερωτήσει προ τον κύριο Σαλανσόν και προ τον κύριο Σαλανκόν και προς τον... και την κυρία Γκόγεν. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Κυρία Μπίλτ, τελευταία στιγμή ε, συζήτησε το λόγο. Ναι, ναι, γιατί θέλω να αφαιρθώ στην ε, συνάδελφο τη Δανία, γιατί και εγώ ασχολήθηκα με τα θέματα αυτά στη Σουηδία. Υπενθυμίζω, δεν ζούμε σε νησιά, ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου οι εναρμονισμένοι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, για την, ε, για την αύξηση του ανταγωνισμού, για τι καλύτερε ε, τιμέ, για περισσότερε επιλογέ των καταναλωτών, όλα αυτά είναι η απάντηση προς του ψηφοφόρου σα. Μία τουλάχιστον Λοιπόν, θα δώσω εμπρεγνώμονε το λόγο πρώτα απ' όλα στον καθηγητή. Και εσύ, όχι, μάλλον και εσείς αν θέλετε να πείτε δύο λόγια, κύριε Σούλτ. Μην ε, νομίζετε ότι σε αποκλείουμε από τη συζήτηση. Εντάξει, όλοι μπορείτε να πάρετε το λόγο. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Και μετά στο τέλος θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Τεστόρη. Σύντομα καταληκτικά σχόλια από τους προσκεκλημένους μας. Λοιπόν, κύριε Αλμάρα πρώτα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ε, ε, αυτό που, αυτό που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σαν πακέτο. Πάντα θα, θα βρείτε παραδείγματα όπου η εθνική σα νομοθεσία μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί. Ε, αλλά θα ήταν λάθο αν αρχίσετε να σχολιάζετε επιμέρου μία-μία τι αλλαγέ. Προσπαθήστε να μεταφέρετε στου ε, ε, ψηφοφόρου σα ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα τη ευρωπαϊκή λύση που προσπαθούμε να βρούμε εδώ. Και να φροντίζετε ότι θα, θα έχουν ε, ε, ότι, ε, και να φροντίσετε ε, να, να, προ, να προστατεύετε τους καταναλωτές σας, αλλά όλες οι πτυχές θα τεθούν στο ύψιστο δυνατό επίπεδο για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ε, και αυτό τελικά είναι το σημαντικό που θα πρέπει να δούμε. Ευχαριστώ. Euh, Ένα σύντομο σχόλιο μετά από το σχόλιο της Ευρωβουλευτή από τη Σκοτία. Ένα από τα καλά της παρουσίασής μου είναι ότι έδειξε ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οδηγία. Υπάρχει σαφέστατη διαφορά μεταξύ κεφαλαίου 3 και κεφαλαίου 4. Στο κεφαλαίο 3 βλέπετε ότι το πράσινο κυριαρχεί, ενώ στο κεφάλαιο 4 έχουμε κυρίως πορτοκαλί, ενδεχομένως και κόκκινο. Άρα, αν ε, δεν θέλετε να ναι, μπορώ να σας πω ότι όντως υπάρχει πρόβλημα για τη Σκοτία γιατί η εγγύηση περνάει από τα πέντε χρόνια στα δύο. Όμως, για την βιομηχανία αυτό που βλέπουμε είναι ότι για την πλήρη εναρμόνιση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, που το τίμημα είναι πολύ ψηλή προστασία για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι η Κομισιόν αυτό το έχει ήδη κάνει για το κεφάλαιο 3, ενδεχομένως να χρειάζεται περισσότερη συζήτηση για το κεφάλαιο 4. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε υπέρ της μικτής προσέγγισης. Θα συμφωνήσω με τον Κάρλος ότι πρέπει να έχουμε μία ανάλυση του πακέτου, όχι να αναφερόμαστε σε διαφορετικές διατάξεις, μία εδώ, μία εκεί. Πρέπει να υπάρξει μία ανάλυση συνολικά του πακέτου. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι ο τίτλος της οδηγίας είναι «Δικαιώματα καταναλωτή», όχι «Δικαιώματα επιχειρήσεων και εμπόρων». Επίσης να πω ότι αν χρειάζεστε οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, η οργάνωσή μου είναι στη διάθεσή σας. Πολύ σύντομα. Ως πρωταθλητές της ε, εσωτερικής αγοράς. Να πω κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί από τις εμπειρίες μας. Οι κάτοικοι του Λοξεμφούργου συχνά ενοχλούνται γιατί τους αρνούνται να τους αποστείλουν προϊόντα ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αυτοί οι ισότοποι ανακαλύπτουν λόγους που έχουν να κάνουν με τον καταγερματισμό των νομικών προϋποθέσεων. Και αυτό δημιουργεί έναν κατακαιρματισμό της αγοράς. Τελικά. Και επειδή πολλοί από εσάς μίλησαν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θεωρώ ότι πολλές ιστοσελίδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων γαλλικές και γερμανικές δεν γνωρίζουν καν τη δυνατότητα τη διασυνοριακή. Οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί επιχειρηματίες σκέφτονται μόνο τη γαλλική ή τη γερμανική αγορά. Άρα δεν έχει μπει η έννοια του διασυνοριακού εμπορίου στο μυαλό τους ακόμη. Αλλά αυτό δεν είναι η βάση της συζήτησης για εμάς. Ευχαριστώ πολύ να αναφερθώ λίγο στο ζήτημα που έδειξε η κυρία Γκέπχαρτε, διαφορά μεταξύ Γερμανίας και Καλλίας. Να πλουστεύσω χοντρικά ε, και να πω ότι κατά δύο ε, πρώτα έτη ε, οι διαφορές σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της επαναχώρησης από, την, από αυτό το συμβόλαιο είναι μικρή. Αλλά από εκεί και μετά μπορεί να υπάρχει μια περίπτωση να υπάρχει ένα δικαίωμα, για παράδειγμα, το οποίο χορηγείται από τις γαλλικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή. Και εδώ δεν θέλουμε να παρέμβουμε, γιατί αυτό είναι και ένα ζήτημα ανταγωνισμού. Αλλά, εάν έχουν περάσει δύο χρόνια και διαπιστωθεί ένα ελάττωμα εκ των υστέρων σε αυτό το προϊόν, η διαφορά σε ό,τι αφορά το δίκαιο είναι τελείω διαφορετική γιατί ουσιαστικά στη Γερμανία εκεί δεν υπάρχουν κανένα είδου δικαιώματα για τον καταναλωτή. Πέρα από κάποιε ορισμένε εξαιρέσει, ενώ στο γαλλικό δίκαιο υπάρχουν εξαιρετικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν ω Γάλλο καταναλωτή, εγώ θα το αναλογιζόμουν πάρα πολύ αν θα πήγαινα στη Γερμανία να αγοράσω κάτι, ένα προϊόν το οποίο έχει ένα σχετικά, μια σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, αν θέλουμε να ε, πραγματοποιήσουμε την ε, κοινή αγορά. Δηλαδή αυτό δεν έχει να κάνει με ή με πολιτισμικές ή οποιασδήποτε άλλες διαφορές, αλλά με διαφορετικές, ε, διαφορετικά δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά την ε, πλήρη εναρμόνιση θεωρώ πως είναι αρκετά υπερβολικά ίσως γενικόλογη η συζήτηση. Δεν μπορούμε να πούμε ε, θα πρέπει να ασχίσει για όλα πλήρης αναρμόνιση ή μερική ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να δούμε ένα προς ένα τους σχετικούς κανόνες, τα σχετικά δικαιώματα. Ε, και ίσως θα πρέπει να εστιάσουμε με αυτόν τον τρόπο τους ώστε να διαπιστώσουμε κάποια σημεία όπως είπε και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία είναι δυνατή η πλήρη αναμόνωση χωρί να χρειάζεται να παρέμβαμε με αυτον τον τροπο του ωστε να διαπιστωσουμε καποια σημεια οπω ειπε και εκπροσωπο τη ευρωπαικη επιτροπη τα οποια ειναι δυνατη η πληρη αναμονωση χωρι να χρειαζεται να παρεύουμε με ιδιαιτερο τροπο στο δικαίωμα του καταναλωτή. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι τομείς οι οποίοι είναι σχετικά απομονωμένοι και ε, στους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε κάτι. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις, ε, την επαναχώρηση, τη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα τη επαναχώρησης και ούτω καθεξής, εκεί θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάτι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σα. Κύριε Σιστόρη, θα ήθελε να μας δώσει κάποια, να κάνει τα καταληκτικά τη σχόλια που δώσω στο λόγο στον κύριο Σφάμπ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω πως ο ε, αγωνιστικός αντίκτυπος ε, ε, της οδηγίας μας στις εθνικές νομοθεσίες, δηλαδή ο πίνακας τον οποίο έχουμε εμβάσει, είναι κάτι το οποίο σας έχουμε παρουσιάσει χωρίς να μας ζητηθεί. Και μπορείτε να τα δείτε και αυτά στη συμφωνία που έχουμε. δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάζουμε πάντοτε το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό και το χθες αντίκτυπο. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε όλα τα προσόντα εντό εισαγωγικών για να το κάνουμε, για να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε όλη την τεχνική επιδομοσύνη. Είναι κάτι το οποίο εμεί ε, προσφέραμε στη συζήτηση. Από εκεί και μετά, α μην είμαστε ντογματικοί ω προ το ζήτημα τη ε, πλήρου εναρμόνιση ή τη ελάχιστη εναρμόνιση. Εμεί θέλουμε να κάνουμε αυτό που είναι υπεύθυνο για τα δικαιώματα του καταναλωτή, δηλαδή βελτίωση τη προστασία των δικαιωμάτων του για όλου του καταναλωτέ σε όλα τα 27 κράτη-μέλη και για τα 480 εκατομμύρια, ε, εκατομμύρια καταναλωτών που κατοικούν σε αυτές. Εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο οδηγεί σε αύξηση της ε, προστασίας, αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή εξετάζουμε πάντα τα δικαιώματα όλων των καταναλωτών. Και απαντώντας ε, συντομία στην κυρία Γκέπχαρτ, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από το Γενικό Ενοχικό Δίκαιο και αυτά δεν εμπίπτουν εδώ στον ε, πεδίο του δικού μας αρμοδιότητων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, όλους ε, πολύ για τις ε, παρεμβάσεις σας και χαρά μου να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας για να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια, να συνοψίσει τη συζήτηση και να μας πει ενδεχομένως ποια θα είναι τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε σε σχέση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να πω πως είμαι πολύ περήφανος ο μέλος αυτής της Επιτροπής, γιατί ενώ άλλες ε, επιτροπές, ε, ε, όπως η Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, οι άλλε ήδη βρισκόνται στη φάση τη ψήφιση. Εμεί ακόμα εξετάζουμε εντελεχώ αυτό το ζήτημα. ακούσαμε μια άποψη που λέει ότι δεν χρειαζόμαστε αυτή την πρόταση γιατί ούτω ή άλλω οι καταναλωτέ λόγω των γλωσσικών εμποδίων και ούτω καθεξής δεν προβαίνουν διασυνοριακά σε αγορέ. Κάτι τέτοιο νομίζω πω μπορούμε από κοινού να το απορρίψουμε γιατί γνωρίζουμε πω υπάρχουν πάρα πολλοί καταναλωτέ οι οποίοι επιθυμούν να αγοράζουν διασυνοριακά. Εγώ για παράδειγμα ήθελα να αγοράσω ένα κράνο σκι ε, ε, αρχές ε, ε, του έτους ε, γιατί και μάλιστα επειδή είχε προκύψει αυτό το ατύχημα ενός γνωστού πολιτικού όταν έκανε σκι είχαν ξεπουληθεί όλα τα κράνη σκι και χρειάστηκε να πάω σε γαλλικό website δηλαδή με τελεία .fr για να μπορέσω να βρω το κράνος μου. Ε, και γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι υπάρχει ένα σουηδική προέλευση ε, ε, κατάστημα το οποίο βρίσκεται εδώ στι Βρυξέλλε και το οποίο δεν προβαίνει σε, δεν, δεν προμηθεύει δηλαδή καταναλωτές στη Γερμανία και αυτό το κάνει πάλι επικαλούμενο τέτοιου είδου διαφορέ. Άρα λοιπόν εγώ είμαι θετικά διατήμενος απέναντι σε αυτή την πρόταση οδηγία, γιατί όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα να προβαίνει οι καταναλωτέ σε περισσότερε δασιονομικές άγορες, αλλά ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να βρούνε και πιο ελκυστικές και πιο φθηνές προσφορές. Όμως ε, θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους εκείνους που πήραν το λόγο και είπαν πως ε, θα είμαστε σε θέση να εναρμονίσουμε το δίκαιο, την ομοθεσία, αλλά δεν μπορούμε ε, εναρμονίσουμε πλήρως την καθημερινή πρακτική σε ό,τι αφορά τη σύναψη των συμβολέων. Ε, δηλαδή εκεί θα συνεχίσουμε να ισχύουν διαφορετικές πρακτικές, παραδόσεις, κουλτούρα, γλώσσα ε, των εκάστοτε κρατών μελών. Το ε, γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια που ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να επιληθεί μόνο με ελάχιστη εναρμόνιση δεν μπορεί να αποτελεί για μας επιχείρημα για να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Εμείς δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ένα βιώσιμο δρόμο, μια βιώσιμη λύση ευρωπαϊκή, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα σε εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την ευρωπαϊκή ε, προοπτική. Ε, νομίζω πως ε, σε αυτό το τομέα είμαστε ουσιαστικά και θα πρέπει να παραμείνουμε εκείνοι που τάσσονται υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής και όταν θα γίνει η πιο τεχνική συζήτηση ε, για αυτή την πρόταση, στα άρθρα 1 έως 3 θα πρέπει να ε, ε, στοχεύουμε προς την πλήρη εναρμόνιση εκεί. Απλά είναι το ζητούμενο βέβαια το πώς θα την επιτύχουμε και τι ακριβώς θα πρέπει να προβλέψουμε. Και ελπίζω πως και ως ε, κοινοβούλιο θα λάβουμε και πιο, πιο σαφή σημειώματα διευκρινιστικά από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά ε, τα δικαιώματα όπω αυτά αναφέρονται τώρα στο κεφάλαιο 4, θα χρειαστούμε περισσότερε διευκρινήσει όπω και αυτέ ζητήθηκαν από τον κύριο Σούλτεν και δηλαδή τι σημαίνει το δικαίωμα αυτό το οποίο ε, ε, τρέχει για δύο ή τέσσερα χρόνια ε, δηλαδή γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις ακόμα και μετά από τρει ημέρες δεν έχει ιδιαίτερο δικαίωμα καθώς ε, σε ε, μηχανήματα πλήρους λειτουργίας να είναι ήδη γνωστό το αν υπάρχει κάτι ή όχι. Άρα λοιπόν εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε να εστιάσουμε σε αυτά που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο, για τον καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το κεφάλαιο 4 βλέπω, διακρίνω κάποια προβλήματα ε, ε, καθώς χρειάζεται εκεί ενδεχομένως ε, να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας στην εθνική νομοθεσία. Είτε συμφωνούμε αυτή όχι. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 5 και τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, στο πλαίσιο του ενοχικού δικαίου, παραμένω εν μέρη αισιόδοξο ότι δηλαδή ε, αυτές οι τρεις, τέσσερις, πέντε προτάσεις θα μπορούσαν να παραμείνουν εκτός επιτροπολογίας ε, και να υιοθετηθούν σε ό,τι αφορά δηλαδή την απόλυτη απαγόρευση στα θέματα των εμπορικών των πρακτικών. Ε, βέβαια κάτι τέτοιο θα πρέπει να συζητηθεί ε, Εντελεχώ με τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα ε, επιτύχουμε να έχουμε μια από κοινού εργασία των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουν το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εργασίες τους. Ελπίζω ε, και πιστεύω πω θα πρέπει ε, να εχουμε μια απο κοινου εργασια των εθνικων εμπειρογνωμονων για να βοηθησουν το συμβουλιο και την ευρωπαικη επιτροπη στι εργασιε του ελπιζω και πιστευω πω θα πρεπει να επιτυχουμε κάτι τέτοιο μόνο με από κοινού συνεργασία, καταλείποντα την εθνική προοπτική και εξετάζοντα λίγο και λαμβάνοντα υπόψη την ε, κοινοτική υπεραξία. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε την τέλεια αγορά, δεν υπάρχει τέλεια αγορά, αλλά μπορούμε ε, να ε, μειώσουμε λίγο τα σφάλματα τα οποία δημιουργούνται και οδηγούν σε στρέβλωση τη αγορά. Πιστεύω λοιπόν πω μπορούμε να τα διορθώσουμε. Παραμένω αισιόδοξο. Σα ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση σήμερα και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα. Uh, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χειροκροτήσατε τους εμπειρογνώμονες, πρέπει να χειροκροτήσετε όλους ε, όσους ε, ήρθαν σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ανδρέας για την διοργάνωση αυτής ε, της ε, ακροάσης. Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις και κάποιες απαντήσεις. Περιμένουμε ακόμη πολλές ε, απαντήσεις και ο εισηγητής μας θα προσπαθήσει να τις βρει τις επόμενες εβδομάδες σε συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές και κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης προκειμένου να καταλήξουμε σε μία πρόταση τροποποιημένη εκ μέρους Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που είδαμε αρκετούς συναδέλφους ε, από την Επιτροπή μας και άλλες ε, και ελπίζω ότι η δέσμευσή σας θα συνεχιστεί. Εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας για σήμερα. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενή μας συνεδρίαση θα είναι την επόμενη Τρίτη από τις 9 μέχρι τις 6.30. Η Αντιπρόεδρος, η κυρία Κόρχολα, θα προεδρεύσει της Επιτροπής όλη την ε, ημέρα, γιατί εγώ θα πρέπει να πάω στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος στο Μάντσεστερ. Θα σας ενημερώσω, θα ενημερώσω μάλλον τους συναδέλφους στο Μάντσεστερ για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Να σας πω ότι το πρωί θα ασχοληθούμε με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα εργασίας. Θα ασχοληθούμε με την προσφορά αερίου και το scoreboard για τους καταναλωτές η κυρία Σάλτεμος ε, θα μπορέσει να μας μιλήσει για τις πληροφορίες στα τρόφιμα. Επίσης ε, θα μιλήσουμε για την εφαρμογή της οδηγίας ε, για την αμοιβή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ενώ τέλος θα έχουμε και μία παρουσίαση για την οδηγία για την οποία μιλήσαμε σήμερα το πρωί, για τις ε, εκδηλώσεις της αγοράς και τέλος, αν σας ενδιαφέρει, μπορούμε να συζητήσουμε για το Solvit, για το εμπόδια για την πλήρη εφαρμογή της ε, εσωτερικής αγοράς και για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις δημόσιες προμήθειες. Για τα τρία αυτά θέματα θα συζητήσουμε το κατά πόσο θέλουμε να κάνουμε έκθεση πρωτοβουλίας. Στο μέλλον θα έχουμε πολύ πλήρη ατζέντα στην Επιτροπή μας, οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές και τους συζητητές και σχεώδεις συζητητές για το έργο τους. Ελπίζω ότι θα σας δώσω την μεθεπόμενη μας συνεδρίαση. Καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Thank you